Eh, Καλημέρα σας. Από τη συνάδελφα. Και φίλοι. Ας ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας, παρακαλώ. Η Επιτροπή των Γυναικών και Ισότητας των Φίλων. Και θα ήθελα καταρχάς να ερωτήσω εάν υπάρχουν προτάσεις για τροποποίηση ή παρατηρήσεις σχετικές με την ημερήσια διάταξη. Αν όχι, ας προχωρήσουμε όπως προβλέπει η ημερήσια διάταξη. Την έχετε λάβει γραπτός. έχετε λάβει ασφαλώς και τα πρακτικά των δύο τελευταίων συνεδριάσεων της 12 η Ιανουαρίου και της 19 9η και 20ης Ιανουαρίου 2009. Εάν δεν έχετε παρατηρήσεις ή σχόλια να καταθέσετε μέχρι το τέλος της συνεδρίασής μας σήμερα, θεωρείτε ότι τα πρακτικά έχουν εγκριθεί. Τώρα ενημερωτικά θα σας πω τα εξή. Έχουμε προβλέψει τη διεξαγωγή μιας δημόσιας ακρόασης για τα πρώτα δύο θέματα στην ημερήσια μας διάταξα. Καταρχάς το κοιτή σε ανωνυμία, ακρόαση δημόσια, η οποία θα μεταδοθεί και μέσω του διαδικτύου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απευθείας και βλέπετε για το απόγευμα. Και έχουμε την κυρία Χάριετ την Βρετανίδα Υπουργό για θέματα οικογένειας και ισότητας. Θα μας ενημερώσει σύντομα για θέματα των γυναικών και ισότητας των ευκαιριών, των ευκαιριών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το απόγευμα προβλέπετε να ψηφίσουμε. Έχουμε μια σειρά εκθέσεων για ψηφοφορία. Και γι' αυτό σας παρακαλώ να φέρετε μαζί σας όλοι την κάρτα σας. Μάλιστα μόλις ενημερώθηκα ότι η εκπομπή της συνεδρίασής μας ήδη έχει ξεκινήσει από το διαδίκτυο. Είμαστε λοιπόν live και γι' αυτό χαμογελάτε. Κρατήστε ένα διαρκές και μόνιμο χαμόγελο στο χείλη γιατί δεν ξέρετε ποια κάμερα θα σας πιάσει και θα μεταδώσει την εικόνα σας ανά τον κόσμο. Αύριο έχουμε μια κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής μας μαζί με την Επιτροπή των Νομικών Υποθέσεων, την Αντιπροσωπεία για το Αφγανιστάν, με θέμα την εισαγωγή δημοκρατικών πρακτικών και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κυρίως των δικαιωμάτων της γυναίκας στο Αφγανιστάν. Όπως ε, και θέματα βασικών ελευθεριών, ισότιμης προσβάσης στον νόμο, Γι' αυτό σας παρακαλώ να είσαστε όλοι και όλες παρόντες αύριο σε αυτή την κοινή συνεδρίαση. Επίσης, την προηγούμενη εβδομάδα έγινε ψηφοφορία για την απαγόρευση των διακρίσεων ε, με βάση το φύλλο για τα θέματα της ισότητας των φύλων, μια πρόταση των πρασίνων. που σε μεγάλο βαθμό είχε περάσει και εγκριθεί και από τη δική μας την Επιτροπή. Στο μέλλον θα πρέπει να αγωνιστούμε και για την αναγνώριση, την ισότιμη αναγνώριση και αυτών που αγωνίζονται για την ισότητα των φύλων και την ισότητα των ευκαιριών. Ευχαριστώ λοιπόν όλους και όλες όσοι ασχοληθήκατε με το θέμα αυτό. Ας προχωρήσουμε λοιπόν τώρα στην ημερήσια μας διάταξη και τη σημαντική συζήτηση που έχουμε για την οδηγία για τη βελτίωση των συνθήκων ε, υγείας και ασφάλειας κατά την εργασία των εγγύων λεχόνων και γαλουχοουσών εργαζομένων. Είχαμε δημόσια συνεδρία, δημόσια ακρόαση στο θέμα αυτό, μάλλον σε ένα συναφέ ζήτημα, ίσως και να θυμάστε ότι είχε κινήσει ενδιαφέρον ιδιαίτερο αυτή η συνεδρία της κυρία Στρέλα συναντήθηκε με τους σκιώδεις εισηγητές και τώρα ήρθε η ώρα να ακούσουμε το έγγραφο εργασίας της. Παρακαλούμε λοιπόν την Αντιπρόεδρο κυρία Στέλλα να λάβει το λόγο. Την ευχαριστούμε ιδιαίτερως για όλη τη δουλειά που έχει κάνει στο θέμα αυτό. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Να ξεκινήσω χαιρετίζοντα την πρωτοβουλία της Κομισιόν για αυτή την πρόταση αναθεώρησης, η οποία είναι πρόσδεκτη και αρκετά εύστοχη. Βεβαίω θα μπορούσε να ήταν πιο φιλόδοξη και να έχει πάει μακρύτερα, ιδίω σε ό,τι αφορά την προώθηση της ενεργούς συμφιλίωσης του επαγγελματικού με τον οικογενειακό βίο, καθώς και με τον ιδιωτικό βίο. Αυτή τη στιγμή, όπως γνωρίζετε, συζητάτε η πρόταση αυτή με τους κοινωνικούς εταίρους, καθώς και αυτή για τις γονικές άδειες, για τις άδειες μητρότητας και πατρότητας. Οι δύο αυτές οδηγίες θα εξεταστούν παράλληλα ώστε να γίνει μια πρόταση συνεπής και συνεκτική που να καλύπτει όλους τους τομείς. Όμως, επειδή δεν υπάρχουν ακόμη ακριβή αποτελέσματα των διαβουλεύσεων των κοινωνικών εταίρων, θεωρώ σημαντικό να διευρυνθεί το πεδίο της οδηγίας αυτής. Για τον επιπλέον λόγο ότι η νομική βάση συνδυασμένη η κοινή νομική βάση επιτρέπει την ε, πρόβλεψη διατάξεων για την προστασία της μητρότητας και της πατότητας ως εξεχουσών κοινωνικών αξιών. Από το χάρτη για την ε, ισότητα που υποβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτού του είδους η συμφιλίωση, αυτού του είδους ο συνδυασμός προκύπτει ως προτεραιότητα εάν ο ρόλος των γονέων δεν βασίζεται στην ε, κατανομή των ευθυνών, ο στόχος συνδυασμού του επαγγελματικού και του οικογενειακού βίου, τόσο για άντρες όσο και για γυναίκες, θα γίνεται όλο και πιο δύσκολη και πιο δύσκολος ο συνδυασμό των δύο. Εφόσον λοιπόν εξετάζουμε το θέμα αυτό στην Επιτροπή μας, πρέπει να θυμόμαστε και το ζήτημα των δημογραφικών ε, δυσκολιών. Έχουμε χαμηλά ποσοστά γενετικότητα στην Ευρώπη, γύρανση του πληθυσμού και γι' αυτό πρέπει να ληφθούν μέτρα τα οποία να αναχαιτήσουν αυτές τις τάσεις. Επίσης να προσθέσω ως έναν επιπλέον λόγο για τη διεύρυνση αυτής της αναθεώρησης οδηγίας, της πρότασης αναθεώρησης ότι κάποιες φορές είναι θύματα στερεοτύπων οι γυναίκες στην κοινωνία και συνεχίζουν να είναι. Δηλαδή τις ε, αντιμετωπίζει η κοινωνία ως μητέρες στον αναπαραγωγικό τους λοιπόν ρόλο και πολύ λιγότερο στον παραγωγικό ρόλο που μπορούν να αναλάβουν θα πρέπει όμως να τις αντιβλέπει κανείς ε, από αυτή τη διτή σκοπιά και ως γυναίκες, μητέρες δηλαδή, αλλά και ως εργαζόμενες που έχουν πλήρη δικαιώματα στο χώρο εργασίας. Θα πρότεινα λοιπόν, όπως άλλωστε προκύπτει και από το εγγραφό εργασίας που σας έχει διανεμηθεί και ήδη μεταφραστεί, θα πρότεινα και θα υποβάλω και μια αναλογή πρόταση για χορήγηση και άδεια ε, πατρότητας μητρότητας ατομική η οποία δεν θα μπορεί να, να μεταβιβαστεί και η οποία θα είναι και αμοιβόμενη για τον σύζυγο, τον σύντροφο της μητέρας, ε, ταυτόχρονα με την άδεια μητρότητας. Επίσης είναι σημαντικό να γίνεται αναφορά και στις περιπτώσεις υιοθεσία. Εκεί θα πρέπει επίσης να αναγνώρισε το δικαίωμα της άδεια, η οποία να κατανείμεται εξίσου μεταξύ των δύο μελών ενός ζεύγους. Σε ό,τι αφορά τη διάρκεια της άδεια πατρότητας, σκοπεύω να προτείνω δύο υποχρεωτικές εβδομάδες και δύο προαιρετικές. Όμως, οι δύο προσωρινές εβδομάδες θα πρέπει και αυτές να αμείβονται κατά ένα ποσοστό 100%. Ως προς την ε, διάρκεια της άδεια μητρότητα, η Επιτροπή προτείνει την ε, επέκταση από 14 σε 18 εβδομάδες. Εγώ πρόκειται να προτείνω 20 εβδομάδες, διότι η Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ισότητα και τις Ίσες Ευκαιρίες μεταξύ άντρων και γυναικών συστήνει παράταση κατά 24 εβδομάδες. Επειδή όμως Προτίθεμαι να προτείνω ούτω ή άλλω την άδεια πατρότητα των δύο υποχρεωτικών και δύο προσωρινών εβδομάδων. Ουσιαστικά δηλαδή τέσσερι συνολικά εβδομάδε, εφόσον ε, εγκριθούν. Γι' αυτό νομίζω ότι αν προτείνω τι 20 εβδομάδε για την άδεια μητρότητα, με τι άλλε 4 της άδεια πατρότητα καταλήγουμε στην ίδια πρόταση με αυτή τη Συμβουλευτική Επιτροπή. Επίση, η Επιτροπή δεν προβλέπει μέτρα για θέματα υγείας δεδομένων των μέτρων του ΠΟΗ, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και των σχετικών ρυθμίσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας, εδώ για, τον... Ε, για αυτή την περίπτωση θα ήθελα να προτείνω τουλάχιστον δύο ημερήσια διαλύματα. Επίσης για την αμοιβή θα πρέπει να είναι, να είναι 100% η αμοιβή, αμοιβόμενη άδεια των γυναικών διότι μπορεί οικονομικώς να πληγούν οι γυναίκες από την απόφαση αυτή να κάνουν παιδιά. Επίσης, η απαγόρευση απόλυσης. Εδώ νομίζουμε ότι η πρόταση της Επιτροπής είναι αρκετά ισορροπή. Όμως τα σχετικά δικαιώματα θα πρέπει να διευρυνθούν και να αφορούν και τον πατέρα, κατά τη διάρκεια της άδειας πατρότητας τουλάχιστον. Έπειτα, για την περίοδο μετά τη διάρκεια, μετά την άδεια μητρότητας. περίοδο κατά την οποία θα πρέπει να προστατεύεται από ενδεχόμενε απολύσει η γυναίκα, η Επιτροπή προτείνει ένα εξάμεινο. Ένα εξάμεινο προστασία μετά την άδεια. Εμείς νομίζουμε ότι η περίοδος αυτή πρέπει να παραταθεί σε 12 μήνες, διότι πολλές φορές οι εργαζόμενοι θα αναγκαστεί να προσαρμοστεί σε μια νέα κατάσταση, σε νέες συνθήκες εργασιακές, κάτι που απαιτεί χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί θα χρειαστεί ενδεχομένως ένα κύκλο κατάρτισης ή και να διοχετευτεί σε κάποιο άλλο κλάδο. Σε ό,τι αφορά την ε, οργάνωση της εργασίας, νομίζω ότι τα δικαιώματα που προβλέπονται για τις γυναίκες θα πρέπει να ισχύουν και για τους άνδρες. Μετά την ε, χρήση της άδειας πατρότητας. διότι είναι περισσότερες οι γυναίκες από ότι οι άνδρες που ανατρέχουν σε αυτό το είδους τα μέτρα ευελιξίας στην ε, οργάνωση της εργασίας, αλλά αυτό προκαλεί έλλειψη ισορροπίας. Και βεβαίως υπάρχουν και αρνητικές συνέπειες. για τις γυναίκες, καθώς και οικονομικό αντίκτυπο για κάποια κράτη-μέλη. Σε ό,τι αφορά την υγεία και την ασφάλεια, εδώ θα πρότεινα τη διεύρυνση του πεδίου εφόσον η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει μόνον να υπάρχει αξιολόγηση των κινδύνων αφότου ενημερώσει για την εγκυμοσύνη της η γυναίκα τον εργοδότη. Γνωρίζουμε όμως ότι οι παράγοντες που προκαλούν αλλά αλλοιώσεις ή γεννητικέ αρωμαλίες που προκαλούν ε, χρωμοσαματικές αλλοιώσεις ή δυσπλασίες ή άλλα προβλήματα μπορεί να ε, αφορούν ε, τις γυναίκες στη φάση αυτή ακριβώς και να επηρεαστεί το έμβριο. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει μια προληπτική προσέγγιση δηλαδή αξιολόγηση επαρκής των κινδύνων στο χώρο εργασίας και αυτό να καλύπτει άνδρες ή γυναίκες σε ηλικία όριμη για αναπαραγωγή. Μπορεί να υπάρχουν χημικές απειλές λόγου χάρη που να ενδέχεται να πλήξουν, να βλάψουν το έμβριο και να αφορούν τον άνδρα ή τη γυναίκα που βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία. ανακεφαλαιώνοντας. Θεωρώ ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία. Η οδηγία αυτή ανάγεται στο 1992. Είναι αρκετά ξεπερασμένη. Έχει αλλάξει πραγματικότητα και οι σύγχρονες ανάγκες. Πρέπει λοιπόν να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία αυτή για να διευρύνουμε το πεδίο της οδηγίας να προβλέψουμε και την άδεια πατρότητας που ούτως ή σε κάποια κράτη-μέλη προβλέπεται και η οποία διαφέρει από την γονική άδεια. Μην προκαλέσουμε σύγχυση δηλαδή μεταξύ της γονικής άδειας και της άδειας μητρότητας ή πατρότητας. Μιλάμε για διαφορετικές έννοιες. Επίσης, κάτι άλλο που ισχυρίστηκε και προέβαλε ως επιχείρημα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε και εμείς ως Επιτροπή και ως Ευρωκοινοβούλιο είναι η σημασία που πρέπει να δοθεί στην συμφιλίωση, στο συνδυασμό μεταξύ επαγγελματικού και οικογενειακού αλλά και ιδιωτικού βίου. Είναι απαραίτητο και οι άνδρες ή πατέρες να εμπλέκονται ευθύ εξ αρχή στην ανατροφή των παιδιών. Γιατί αυτό δεν είναι δικαίωμα μόνο των ενηλίκων, αλλά θα πρέπει να έχουν και τα παιδιά το δικαίωμα να υπολογίζουν όχι μόνο στην παρουσία και τη συμμετοχή της μητέρας, αλλά και του πατέρα στην ανατροφή τους. Για την ε, καλή υγεία ενός παιδιού αυτό είναι απαραίτητο. Τα δικαιώματα των, ενός πατέρα στην ανατροφή του παιδιού του είναι σημαντικά. Αυτό είναι και ο ρόλο λοιπόν τη άδεια πατρότητα και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που όλοι το ευχόμαστε και το επιδιώκουμε και ελπίζω οι συνάδελφοι τη Επιτροπή να στηρίξουν την πρότασή μου. Όπω είπα, η κοινή νομική βάση μα επιτρέπει αυτού του είδου την διεύρυνση του πεδίου τη οδηγία. Η προηγούμενη οδηγία έλεγε απλώς ότι πρέπει να προστατεύεται η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων. Όμως, εδώ η συμπερίληψη στο 3 του άρθρου 143 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής, των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που μιλάει για την προώθηση της ισότητας και των ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών, αυτό επιτρέπει κατά την άποψή μου και κατά την άποψη των νομικών εμπειρογνωμόνων με τους οποίους μπόρεσα να ανταλλάξω απόψεις, αυτό επιτρέπει λοιπόν ακριβώς τη διεύρυνση του πεδίου διεύρυνση που τη βρίσκω πολύ θετική. Περισσότερο μάλιστα από ότι η διεύρυνση προκειμένου να παραταθεί η διάρκεια της άδειας μετρότητας. Θέλουμε να υπάρχει νομίζω κατανομή των ευθυνών μεταξύ άνδρων και γυναικών ούτω ή Είναι κάτι που το επιδιώκουμε. Οι άνδρες και γυναίκες να μοιράζονται τις ευθύνε και στο δημόσιο βίο και στο ιδιωτικό. Αυτό νομίζω ότι ούτω ή άλλω ανταποκρίνεται και στο στόχο τη στρατηγική τη Λισαβόνα. Ακριβώ για αυτού του λόγου λοιπόν θεωρώ ότι είναι άκρα σημασία η διεύρυνση αυτή τη οδηγία ώστε να συμπεριληφθεί και η άδεια πατρότητας. Νομίζω ότι η διεύρυνση λοιπόν αυτή είναι σημαντική. Τέσσερις εβδομάδες μέγιστη διάρκεια. Δύο υποχρεωτικές εβδομάδες όπως σας είπα και δύο προαιρετικές. Πρέπει να αλλάξουν και οι νεοτροπίες. Αυτό είναι σημαντικό. Μας λέει η εμπειρία μας ότι σε χώρε που έχει προβλεφθεί άδεια πατρότητας αρχικά χρησιμοποιήθηκαν περιορισμένα, σε μικρό βαθμό από τους άνδρες, λόγω των στερεοτύπων, λόγω των προκαταλήψεων. Όμως, σταδιακά, σιγά σιγά προσαρμόστηκαν και οι άνδρες, ξεπέρασαν αυτού του είδους τις δυσκολίες και σήμερα τα αποτελέσματα είναι αρκετά ενθαρρυντικά. Η χρήση της άδεια πατρότητας αυξάνεται χρόνο με το χρόνο στα κάτι μέλη όπου προβλέπεται ως δικαίωμα. Έχετε στα χέρια σας, συνάδελφοι, το έγγραφο εργασία. Εκεί εκφράζονται οι σημαντικότερες ε, γραμμές και προτάσεις της δικής μου δουλειάς για την πρόταση αναθεώρηση της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εδώ όλες σας οι προτάσεις, όλες σας οι συμβουλές για να βελτιωθεί η πρόταση αυτή είναι καλοδεχούμενες. Θέλουμε να εγκρίνουμε ένα έγγραφο που ακριβώ να ανταποκρίνεται στι ανάγκε των γυναικών και να ευνοεί και την ε, ισότητα καθώ και τι ίσες ευκαιρίε μεταξύ των δύο φύλων. Ευχαριστώ. Ε, Σας ευχαριστούμε πολύ, λέει η πρόεδρο προ την εισηγήτρια. Τώρα, να δώσουμε το λόγο τους συναδέλφους. Κυρία Πέτρα, πρώτη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Συγχαρητήρια στη συνάδελφα για την έκθεσή της. Το έχει πολύ ζυγίσει, είναι πολύ τολμηρά τα όσα διατυπώνει και θεωρώ ότι τώρα που κοντιάζουμε το πρόβλημα αυτό σοβεί αυτή η κρίση που έχει το συνέπειε στη ζωή μας. Όμως νομίζω ότι για το θέμα προκειμένου είναι συνθήκες ευνοϊκές. σύμφωνα με τις προτάσεις όπως διατυπώθηκαν, Φερρυπίν ε, όσον αφορά τη διάρκεια. Α, τη διάρκεια της ε, άδειας μητρότητας, η οποία θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να ε, παρατείνεται στην Ρουμανία. Ξέρετε ότι έχουμε προβλήματα σχετικά με αυτό. Ε, και προβλέπεται μια διαμητρότητα διετής κάτι το οποίο μας δίνει μια όθηση για αυτή την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επίσης συμφωνώ με την ε, άλλη πρόταση Ότι δηλαδή με την έκθεση αυτή δίνουμε μια απάντηση και στην πρόκληση του δημογραφικού γιατί κατά αυτόν τον τρόπο θα θα, θα, θα βοηθήσουμε τον υπάρχει καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικού και οικογενειακού βίου. Επίση, και αυτό πρέπει να γίνει και για αυτού του πρώτου μήνε τη ζωή του ανηλίκου, του παιδιού, είναι πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά την ορθή απάντηση σωματική, ψυχολογική, πνευματική. Σύμφωνα επίση και με την πρόταση που διατυπώθηκε όσον αφορά την, ε, τις ρυθμίσεις σχετικές με τις απολύσεις. πολύ αξιόλογη η έκθεση, πολύ ποιοτική και επίσης θα πρέπει να σας πω για άλλη μια φορά ότι συμφωνώ με όλες τις και σας ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε κυρία Πέτρε. Κύριε Κοτάρτη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Και εγώ Θέλω να ευχαριστήσω την Αντιτέ Στρέλα και για το έγγραφο που μας υπέβαλε και για τις προτάσεις της γιατί και εγώ συμμερίζομαι την σημασία την έμφαση που έχει δώσει στο να προβλεφθούν νέες προοπτικές ό,τι αφορά την υιοθεσία, την αδιαπατρότητας, τις πτυχές που έχουν να κάνουν με την ευελιξία είτε πριν είτε κατόπιν όταν πρέπει να ληφθεί υπόψη είτε η κατάσταση της εργαζόμενης μητέρας ή το τι συνέπειες μπορεί να έχει γέννηση ενός βρέφους ή υιοθεσία ενός μωρού. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι υπάρχουν αλλαγές αλλαγές τις οποίες δεν μπορούμε πλέον να μην λαμβάνουμε υπόψη. Δεν είμαστε στο 1992 και έχουν αλλάξει τα πράγματα. Η αλλαγή που έχει συμβεί είναι μεγάλη. Δεν μιλάμε για μία απλή εξέλιξη. Μιλάμε για κάτι που έχει προσθεθεί στις προηγούμενες καταστάσεις. Δηλαδή, πέρα από την προστασία της εργαζόμενης μητέρας, Τώρα πρέπει να φροντίσουμε προστασία αυτή να διευρυνθεί και να καλύψει και το ίδιο το παιδί. Να δούμε δηλαδή ποιε είναι οι απαιτήσει και ανάγκε του παιδιού συμπεριλαμβανομένου του παιδιού που έχει υιοθετηθεί, που το έχουν εμπιστευτεί σε ένα ζεύγο. Και εδώ πρέπει να καλυφθεί και ο ρόλο του πατέρα. Δεν λέμε να περάσουμε από την προστασία τη μητέρα στην προστασία του τέκνου, αλλά να προσθέσουμε την προστασία του παιδιού. Μέχρι τώρα επικεντρωνόμασταν μόνο στην ε, προστασία των της μητέρας. Τώρα θα πρέπει να συνοδεύσουμε και να λάβουμε υπόψη και την μέρημνα για το παιδί. Θα συμφωνήσω λοιπόν εδώ με την εισηγήτρια και μετά όσα διάβασα στην έκθεσή της και θα προσέθετα στα σχόλιά μου αυτή τη στιγμή δύο πράγματα. Πρώτον, <clears throat> νομίζω ότι στην επιχειρηματολογία μας κάπου θα πρέπει να ακουστεί ως θέση από την πλευρά μας ότι δεν συμφωνούμε σε όλα τα επιχειρήματα σε όλε τι απόψει τη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όταν λέει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι προτείνει να περάσουμε από 14 σε 18 εβδομάδε, εδώ πιστεύω ότι βασίζεται σε απόψει αρκετά αρνητικέ. Διότι θεωρεί ότι αυτό ως διάρκεια επιτρέπει την ενίσχυση του δεσμού μεταξύ μητέρα και παιδιού. Τέσσερι εβδομάδε πιστεύω και εγώ είναι σαφώ χρήσιμε. Αλλά α παραδεχτούμε και α είμαστε ειλικρινεί μεταξύ μα ότι δεν αλλάζουν και πλήρω το δεσμό μεταξύ μητέρα και τέκνου. Ενισχύεται εν μέρει ο δεσμό αυτό, αλλά δεν αρκεί. Και το επικίνδυνο εδώ είναι ότι σε δύο σημεία λέει το κείμενο τη Κομισιόν ότι η παράταση τη διάρκεια τη άδεια μητρότητα επιτρέπει να φανταστούμε ότι έτσι καλύπτεται και απορροφάται και η γονική άδεια. Άλλο όμως είναι η άδεια μητρότητας, άλλο η άδεια πατρότητας και άλλο η γονική. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπονοεί ότι με την παράταση της άδεια ματρότητας λόγου χάρη οι εταιρείε θα έχουν λιγότερα προβλήματα όταν γίνεται αίτηση για γονική άδεια. Ε, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα γιατί υπάρχει σύγχυση μεταξύ των δύο και θα πρέπει να το επισημάνουμε κατά κάποιο τρόπο, ότι το, εντοπίσαμε αυτό και ότι είμαστε καθέτως αντίθετοι. Το δεύτερο σημείο που θα ήθελα να επισημάνω αφορά την προστασία και την ασφάλεια της εργαζόμενης γυναίκας. Θα επανέλθω σε αυτό. Νομίζω ότι ακριβώς ε, στο διάστημα από το 92 σήμερα θα πρέπει να γίνει ακόμα ένας συσχετισμός όχι μόνον σε ό,τι αφορά τη, τους κανόνες και τις διατάξεις για τις γονικές άδειες ή τη συμφιλίωση επαγγελματικού και οικογενειακού με ιδιωτικό βίο, αλλά και σε σχετισμό με το ωράριο εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά λόγου χάρη, αλλά όχι και αποκλειστικά, σε ό,τι αφορά την νυχτερινή εργασία των γυναικών. Διότι εδώ οι πτυχέ ασφάλεια και υγεία των γυναικών που εργάζονται τη νύχτα είναι ιδιαίτερε. Υπάρχει ένα πρόβλημα σε κάποιε χώρε μάλιστα, όπου προβλέπεται απαγόρευση τη νυχτερινή εργασία των γυναικών λόγω της ε, περίοδου αυτής της μητρότητα, δηλαδή και τη εγκυμοσύνη και των πρώτων μηνών τη μητρότητα. Θεωρώ αλλά αυτό είναι μια συζήτηση που ενδεχομένω να πρέπει να κάνουμε μεταξύ μα. Θεωρώ ότι εδώ, το θέμα είναι να προστατευτεί η ασφάλεια και η υγεία των γυναικών. Και θα πρέπει να επιδιώξουμε να προβλεφθεί μια πρόταση, μια σκέψη, ένα σχόλιο από τη δική μας την πλευρά, ώστε να εντοπίσουμε πώ οι δικέ μα θέσει για την υγεία και την ασφάλεια των γενικών την περίοδο αυτή θα συσχετιστούν και με την οδηγία για το ωράριο εργασία. Ιδίω, όπω προείπα, ό,τι αφορά την απαγόρευση τη νυχτερινή εργασία. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε κύριε Κοτάρτη, λέει η πρόεδρος. Και τώρα έχει το λόγο η κυρία Φιγκερέντο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα συμφωνήσω με πολλά από τα σημεία που σχολιάστηκαν προηγουμένως σε σχέση με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι μια πρόταση που την περιμέναμε γιατί είναι πραγματικά ξεπερασμένη η προηγούμενη οδηγία όμως τελικά δεν ανταποκρίνεται στις προσδικίες μας. Δεν ανταποκρίνεται σε αυτά που επιθυμούσαμε αυτή τη στιγμή. Διότι θέλαμε να έχουμε μια προσέγγιση πολύ ευρύτερη και για τους λόγους που ανέφερε η κυρία Γκοτάρντι. Χρειάζεται εδώ μια άλλη προσέγγιση, μια άλλη προοπτική, όχι μόνο για να περασπιστούμε τα δικαιώματα των γυναικών πλέον, αλλά και των παιδιών. Αυτό προϋποθέτει μια ευρύτερη θεώρηση του θέματος. Η διάρκεια της άδειας μητρότητας ή ο θυλασμός μπορεί να επηρεάσουν τα μοντέλα εργασίας, τα ωράρια εργασίας πλέον. Επίσης η άδεια πατρότητας είναι μέρη αυτής της ευρύτερης θεώρησης. Οπότε τέτοια συζήτηση και εξέταση του θέματος θα πρέπει να γίνει κιόλα. Και εδώ είναι θέμα, ένα θέμα ότι από την πλευρά πολλών επιχειρήσεων δεν ε, πληρούνται υποχρεώσεις και η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται συνεχώς, ιδίως στην Πορτογαλία, δεν ε, πληρούνται όλες οι υποχρεώσεις έναντι των γυναικών. Ε, ήδη την εβδομάδα αυτή συναντήθηκα με γυναίκες κάποιων επαγγελματικών κλάδων, κλάδων που, μου έλεγαν ότι υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κατηγοριοποιηθεί ως εταιρείε κοινωνικής ευθύνες. Και μάλιστα ε, περικόπτουν την περίοδο φυλασμού λόγου χάρη ή θέλουν να καταργηθούν τελείως ή λαμβάνεται τελείως διαφορετικά υπόψη το θέμα των γυναικών που μπορεί να είναι χείρες ή μόνες με παιδιά. Μας λένε ότι δεν έχουν που να αφήσουν τα παιδιά τους. Και οι επεύθυνοι, οι προϊστάμενοι των επιχειρήσεων, στις επιχειρήσεις τους, τους λένε τι να σας κάνουμε, βρείτε μια λύση, ή αφήστε τη δουλειά σας, φύγετε. Αυτό λοιπόν είναι σημαντικό για να μην ξεχνάμε ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχουν κάποιοι όμιλοι όπως ο ΣΑΝ που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως όμιλοι κοινωνικής ευθύνης λόγου χάρη. Άρα ο στόχο δεν είναι μόνο να διαβρύνουμε τα δικαιώματα που προβλέπονται, αλλά να υποχρεώσουμε και αυτού που να τα χορηγούν ε, να, τα, ε, να πληρώνουν τι υποχρεώσει του. Κάτι που σήμερα δεν γίνεται. Δεν υπάρχει απαραίτητο υλοποίηση. Ιδίω στην Πορτογαλία, όπω σα είπα, υπάρχουν φορεί, υπάρχουν δημόσιες, ε, δημόσιοι φορεί που είναι ακριβώ υπεύθυνοι για την εφαρμογή τη νομοθεσία και δεν πληρώνουν τι υποχρεώσει του. Δεν αρκεί λοιπόν. Δεν αρκεί να κάνουμε νέε προτάσει μόνον. Αυτό νομίζω είναι σημαντικό, το επαναλαμβάνω. Χρειαζόμαστε ε, να δούμε τι μέτρα θα λάβουμε για να εκτελεστούν αυτά που ήδη προβλέπονται. Δεν μπορούμε να επιτρέπουμε το να εξακολουθούν καταστάσεις όπως αυτές που σας προανέφερα και που άκουσα να μου αναφέρουν γυναίκε από πολλούς επαγγελματικού κλάδους. Τώρα πρόσφατα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Φιγκερέντο. Κυρία Μπάουερ, ευχαριστώ πολύ. Οι δηλώσει των συναδελφών με αφού <clears throat> να λάβω και εγώ το λόγο, να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Βεβαίω, η βελτίωση των δικαιωμάτων στον τομέα αυτό είναι αναπόφευκτη. Και θα έλεγα επίση ότι όταν υπάρχουν ε, χώρες με πολύ πιο μακρά περίοδο ε, άδειας μητρότητας οι πιο αυστηρούς κανόνες που προστατεύουν ε, από την εκτερινή εργασία ή από άλλες ε, δύσκολες συνθήκες της ε, μητέρες. Θα πρέπει με πολύ μεγάλη προσοχή να τις εξετάσουμε. Πρέπει όμως να επισημάνουμε ότι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε μια μεμονωμένη προσπάθεια γιατί υπάρχει ολόκληρο πλέγμα κανόνων και διατάξεων που προστατεύουν την μητέρα στο χώρο εργασίας Πρόκειται για κανόνες πολλέ φορέ δεν υπάγονται νομοτεχνικά στη γενική νομοθεσία, αλλά απλώ εφαρμόζονται με κάποιο διάταγμα και ίσω για αυτό το λόγο λανθάνουν τις προσοχή μας, αλλά υπάρχουν. Βέβαια το ζητούμενο είναι ποιο θα καταβάλει τα έξοδα, το κόστο αυτών των ε, κανόνων, γιατί για να, για να δεχθούμε έναν τέτοιο κανόνα θα πρέπει να ξέρουμε τι είδους επιπτώσεις θα έχει. Όταν βλέπουμε οι τράπεζες να ε, σώζονται, να βάζει το κράτος ε, βατέ το χέρι στη τσέπη για να σώσει τις ε, τράπεζες από την κρίση που αντιμετωπίζουν, ίσως πρέπει να αναλογιστούμε ότι τα προβλήματα είναι πολύ πιο περίπλοκα. Και άρα τα προβλήματα αυτά, τα κοινωνικά, τα οικονομικά δεν μπορούμε να τα παραγνωρίσουμε και θα πρέπει ίσως να κάνουμε μια αναφορά σε αυτά. Γιατί με την επιβολή τέτοιου είδου υποχρεώσεων επιβαρύνονται ιδιαίτερα οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις συνεπάγεται αυτό σημαντικό κόστος για μια τέτοια επιχείρηση. Άρα θα πρέπει να βρούμε κάποιες λύσεις για αυτές. Δεν αρκεί να κάνουμε, να εισάγουμε την νομοθεσία χωρίς να αναλογιζόμαστε τις συνέπειες, γιατί βέβαια θα βρεθεί ο τρόπος να αντιπαρέλθουν τελικά την ε, νομοθεσία, να την καταστρατηγήσουν και να μην την εφαρμόσουν. Όπως είπε και η κυρία Φεγγερέντο, θα πρέπει να βρούμε κάποιες ε, λύσεις ρεαλιστικές. Επίσης θα πρέπει να φροντίσουμε να εισαγάγουμε και κυρώσεις ως προς την, ε, το ενδεχόμενο της παράβασης ε, των καρών αυτών. Φερρυπίν. Ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει μια αποζημίωση. Η μητέρα η οποία δεν τη λαμβάνει αναγκάζεται να καταφύγει στα δικαστήρια. Ε, αυτό βέβαια σημαίνει ένα επιπλέον κόστος. και ναι μεν υπάρχει λύση της δικαστικής ε, αντιμετώπιση των προβλημάτων, αλλά όταν ένα κράτος δεν θέλει να εφαρμόσει τους κανόνες, απλώς δεν θα τους εφαρμόσει. Άρα θα πρέπει να φροντίσουμε να επιβάλλουμε και κυρώσεις σε εκείνους, σε εκείνα τα κράτη που δεν το πράττουν και οι εργοδότες οι οποίοι δεν εφαρμόσουν σωστά την νομοθεσία θα έπρεπε ενδεχομένως να αποκλειστούν από την κοινωτική χρηματοδότηση. Η δική μου εμπειρία από την προηγούμενη έκθεση, η δική μου εμπειρία και από τη δουλειά που έχω τα τελευταία 7 χρόνια στην Επιτροπή μας, μου δείχνει ότι δεν είμαστε αρκετά αποτελεσματικοί ε, στην νομοθεσία που εισάγουμε, γιατί δεν προβλέπονται οι απαραίτητες κυρώσεις. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Μπάουερ. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο παρακαλώ να λάβει το λόγο μέσω των εκπροσώπων τους. Κυρία Μπανκέρ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την συγγήτρια και, τις, ε, και για τις τέτοιες σημαντικές της παρατηρήσεις. Φυσικά δεν είμαι σε θέση να σας δώσω τώρα την ε, οριστική θέση της Επιτροπής για τις ε, παρατηρήσεις αυτές που αφορούν την πρότασή μας, αλλά μια πρώτη απάντηση με αντιδράσεις που μπορώ να κατανείμω σε δύο κατηγορίες μπορώ να δώσω. Πρώτον, η συγγήτρια και ορθά υπογραμμίζει τις ευθύνες που καλούνται να αναλάβουν οι πατέρες στα οικογενειακά βάρη. Αυτή είναι μια πάγια θέση άλλωστε και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όταν μιλούμε δηλαδή για συμφιλίωση, εμείς εννοούμε πάντοτε όχι μόνο τη γυναίκα, αλλά και τη γυναίκα και τον άντρα. Εννοούμε άλλωστε ισότιμες ευκαιρίες μεταξύ ανδρών και γυναικών. Παγίως επίσης ακολουθούμε στις εργασίες μας τον στόχο αυτό και εδώ θα ήθελα να αναφερθώ και στις διαβουλεύσεις που ξεκινήσαμε με τους κοινωνικούς εταίρους ως προς το θέμα της συμφιλίωσης η οποία διαβούλευση, οι οποίες διαβουλεύσεις εν τέλει οδήγησαν ε, στη Συμφωνία των Κοινωνικών Εταίρων για τη μεταρρύθμιση της οδηγίας περιγονικής άδειας. Επίσης άτυπες διαβουλεύσεις που ξεκινήσαμε δυνάμει του άρθρου 138 της συνθήκης, όπου ιδιαίτερα υπογραμμίστηκε ο στόχος της διευκόλυνσης και της ε, παροχής ε, κινήτρων προς τον πατέρα, ώστε αυτός να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο από τα οικογενειακά βάρη. Επίσης, ε, συμφιλίωση αλλά και περισσότερες ευθύνες για τον πατέρα καταγράφονται στην, στο φύλλο πορείας για το 2006-2006 που δημοσιεύτηκε το 2006. Άρα είμαστε σύμφωνοι με το στόχο αυτόν, να ενθαρρύνουμε τον πατέρα περισσότερο και να καταλήξουμε τελικά στην κατάσταση αυτή κατά την οποία θα υπάρχει πιο ισόρροπη κατανομή των ρόλων μεταξύ του πατέρα και της μητέρας στην ανάληψη των οικογενειακών ευθυνών. Τούτου λεχθέντος βέβαια πρέπει να δούμε ότι εδώ η μεταρρύθμιση είναι μόνο ένα τμήμα των προτάσεων, της δέσμης προτάσεων που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2008 παράλληλα και με μια έκθεση για τις ε, ε, υποδομές περί για τα παιδιά μέσα στο πλαίσιο και της ε, πορείας της την οποία θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική και επίση υιοθετήσαμε προτάσει για την υποστήριξη των συζύγων που θα συζητήσει αργότερα η Επιτροπή σα. Έχουμε επίση ενεξελίξει τις διαπραγματεύσεις μεταξύ κοινωνικών εταίρων για την μεταρρύθμιση τη ε, οδηγία περί γονική άδειας και εμεί νομίζουμε ότι θα έπρεπε να εισαχθεί και η δυνατότητα τη άδεια, τη γονική σε περίπτωση υιοθεσία και η εισαγωγή της γονικής άδειας για τον πατέρα και όχι για την περίπτωση μόνο του τοκετού. Όπως ξέρετε η άδεια τοκετού υιοθετήθηκε εισήχθη ως μέτρο εδώ και 15 χρόνια. Πρέπει να εξυγχρονιστεί το νομοθέτημα αυτό, κατά την άποψή μας όμως, είναι ένα νομοθέτημα το οποίο πάνω απ' όλα απευθύνεται στη γυναίκα. Στόχο έχει τη διαφύλαξη της υγείας και ασφάλειας της εγγύου και της ε, Λεχώνας. Άρα λοιπόν κύριος στόχος του είναι η γυναίκα όπως είπα, ενώ η άδεια για τον πατέρα, η γονική, η σχετική με την οικογένεια άδεια με τον πατέρα θα πρέπει να ενταχθεί περισσότερο στην οδηγία περί γονικής άδειας. Άλλο ένα σημείο που ακούστηκε κατά τη συζήτηση και στο οποίο θα θέλω να αναφερθώ είναι το εξή. Δεν νομίζω ότι αναμειγνύεται εδώ η άδεια το κετούμε με την αγωνική άδεια. Άλλωστε στην επιχειρηματολογία μας εξηγούμε γιατί θέλουμε ε, η άδεια το κοιτού να παραταθεί από τις 14 στις 18 εβδομάδες. Πρώτος λόγος βέβαια είναι η υγεία και η ασφάλεια της μητέρας, αλλά και η δυνατότητα που θέλουμε να της προσφέρουμε να μείνει πιο κοντά στο παιδί της, πιο πολύ καιρό κοντά στο παιδί της, να θυλάσει, να αναπτύξει γερούς και υγιείς δεσμούς με το παιδί της που θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικού. Βέβαια, οι τέσσερι ίσω επιπλέον εβδομάδε μπορεί να μην σημαίνουν μια ριζική αλλαγή, πλην όμω είναι σημαντική αλλαγή και πάνω απ' όλα ένα βήμα προς την ορθή κατεύθυνση. Για δε τη γονική άδεια, δεν λέμε ότι θα πρέπει οι γυναίκες πια να αξιοποιούν τη γονική άδεια, αλλά πάνω απ' όλα λέμε ότι όταν ένα παιδί είναι ηλικίε 18 εβδομάδων, ίσως η μητέρα είναι καλύτερα σε θέση, ευχερέστερα σε θέση να βρει την κατάλληλη μέρημνα υποδοχή για το παιδί, παρά όταν το παιδί βέβαια είναι 14 εβδομάδων, όταν είναι πιο μικρό. Αυτό είναι το επιχείρημά μας για τη γονική άδεια, ότι είναι πιο εύκολο να βρεθεί η υποδομή μέρημνας για το παιδί 18 εβδομάδες μετά το τοκετό. Και άρα μπορεί τη γονική άδεια η μητέρα να την αξιοποιήσει σε ένα μεταγενέστερο στάδιο της ζωής του παιδιού της. Αυτά είχα να πω προς το παρόν. Ευχαριστώ ιδιαίτερα την εισηγήτρια Και βέβαια με χαρά θα συνεργαστώ μαζί σας πάνω στην πρόταση αυτή. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα επιτρέψτε μου να ζητήσω, το λόγο, να, ζητήσω να λάβει το λόγο και ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για όλα αυτά τα οποία μας εξέθεσε για την πρότασή της. Ήθελα να σας πω εγώ Συμβουλίου τα εξής. Ε, βρισκόμαστε ακόμα σε πρώιμο στάδιο όσον αφορά την προβληματική και επίσης οι διαπραγματεύσεις όπως γνωρίζετε άρχισαν τώρα με την Γαλλική Προεδρία. Οπότε συνεχίζουμε τις διαβουλεύσεις με την Τσεχική Προεδρία και θεωρούμε ότι πρόκειται πάντως για ύψιστη προτεραιότητα. Είναι κάτι το οποίο αφορά την κοινωνική πολιτική. Και επομένως θα συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση και κατά την Τσεχική Προεδρία. Έχουμε συγκροτήσει μια ομάδα εργασίας έχει συναντηθεί μόνο μία φορά. Όμως κατά την επόμενη πολιτική Σύνοδο ε, θα έχουμε και άλλη μία συνεδρίαση αυτής της ομάδας εργασίας. Τώρα προσπαθούμε να κάνουμε μία ανάλυση του σχεδίου της οδηγίας και ιδίως ασχολούμεθα με τα θέματα που ενδιαφέρουν περισσότερο τα κράτη-μέλη από το σχέδιο κειμένου. Πάντως μέχρι σήμερα έχει συζητηθεί όπως είπαμε αυτή, αυτό το κείμενο και τώρα συζητούμε το άρθρο 8 το οποίο ακριβώς αφορά την διάρκεια της ε, μητρικής αδείας. Θεωρούμε ότι μέσω αυτού του άρθρου θα έχουμε τις πιο εντυπωσιακές αλλαγές σε σχέση με την οδηγία του 92. σώματα εργασίας. Συζητήσαμε θα το άρθρο 8, το κάθε κατασμένο φυσικά έχει διαφορετική γνώμη. Και φυσικά υπάρχει και θέμα ε, απόκλησης των εθνικών νομοθεσιών και είναι πάρα πολύ δύσκολο βέβαια το να μπορέσουμε να συγκεράσουμε αυτές τις απόψεις. Πάντως θα κάνει ό,τι μπορεί η Τσεχική Προεδρία ούτως ώστε να συνδυάσουμε αυτές τις διαφορετικές απόψεις των κρατών μελών. Και έτσι, όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδρομή, να έχουμε κάποια και οποιαστά αποτελέσματα και να μπορέσουμε να έχουμε καταλήξει σε κάποια συνένεση. Επίσης, οφείλω να σας πω ότι στην Ιερνή Σύνοδο ή στο Συμβούλιο που θα γίνει το Μάρτιο και αυτό πρόκειται να συζητηθεί, έχουμε εκπονήσει ε, κάποια έγγραφα για τους υπουργούς για να γίνει ανταλλαγή απόψεων οπότε αυτή η συζήτηση που θα γίνει από τους υπουργού νομίζω ότι πρόκειται να δείξει την κατεύθυνση από τα πράγματα στο μέλλον σε σχέση με το σχέδιο οδηγίας. Βεβαίως και πρόκειται να συνεργαστούμε με βουλευτές, με τον εισηγητή και έτσι να μπορέσουμε η θέση του ε, Κοινοβουλίου να προσεγγίσει όσο γίνεται τη δική μας. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Εμείς σας ευχαριστούμε, λέει η Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε για όλα αυτά τα οποία μας εξηγήσατε. Τώρα, νομίζω ότι θα πρέπει να δευτερολογήσει η συγγήτρια. Ευχαριστώ, Πρόεδρο. Να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τις συνεισφορές τους, τα σχόλια, τη συμβολή τους, για την αποτίμηση των δικών μου των προτάσεων και ήθελα εδώ να δώσω κι εγώ κάποιες τελικές μου σκέψεις. Εδώ μιλάμε για μια οδηγία που εφόσον θα πρέπει να μεταφερθεί στι εθνικέ νομοθεσίε, θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα κοινό παρονομαστή που να ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό δεν απαγορεύει, το προβλέπει άλλωστε η οδηγία. Τα κράτη-μέλη όπου έχουν πιο ευνοϊκή νομοθεσία να μπορούν να συνεχίσουν να την εφαρμόζουν. Γνωρίζουμε ότι η κατάσταση διαφέρει πολύ από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. ιδίω ό,τι αφορά τη διάρκεια, αλλά και την αμοιβή. Δηλαδή υπάρχουν κράτη-μέλη που προβλέπουν την ελάχιστη διάρκεια για την άδεια μετρότητας των 14, 14 εβδομάδων και υπάρχουν και κάτι μέλη που προβλέπουν τη διάρκεια του 52 βάσει τη οδηγία 92-85. Έτσι λοιπόν είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα όσο ότι αφορά και την ε, πληρωμή. 100% αμοιβή για κατά την άδεια τη διάρκεια σε κάποια κάτι μέλη, ενώ σε κάποια άλλα 100% για ένα διάστημα και μετά κάποιο είδου ε, επιδότηση, επιχορήγηση. Ε, καταστάσεις δηλαδή πολύ διαφορετικές μεταξύ τους. Τώρα για τα σχόλια των συναδέλφων να πω το εξής. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή θα ήταν καλό να διευρύνουμε υπερβολικά την όλη έννοια της άδειας μητρότητας. Διότι εντοπίζουν οι μελέτες ότι και η παρατεταμένη απουσία της γυναίκας από τον εργασιακό χώρο μπορεί να είναι πολύ επιζήμια. Και δεν υπάρχουν και ειδικά ωφέλη από ένα συγκεκριμένο διάστημα και μετά και για το παιδί. Δηλαδή είναι οι πρώτοι μήνες που είναι καθοριστικοί. Αυτή ναι, γιατί υπάρχει ο συναισθηματικός δεσμός, στην συναισθηματική σχέση του παιδιού με την ε, μητέρα. Το δέσιμο. Ε, έπειτα τα πλεονεκτήματα είναι σχετικό αν είναι περισσότερα από τα μειονεκτήματα. Και υπάρχουν και προκαταλήψεις που λένε ότι είναι πιο επικίνδυνο, πιο απειλητικό να προσλάβει κάποια γυναίκα από έναν άντρα, γιατί μπορεί να φύγει με άδεια εγκυμοσύνης. Αυτό θα, θα βλάψει ακόμη περισσότερο τις γυναίκες, εάν δεν βρίνουμε πάρα πολύ την όλη έννοια της άδειας μητρότητας. Επίσης, σε ό,τι αφορά την νυχτερινή εργασία ή ε, τις ώρες τις υπερορίες, εδώ θα πρέπει να αφήσουμε κάποια ευελιξία. Κάποιο περιθώριο ευελιξίας. Δηλαδή, εάν οι εργαζόμενοι Ε, εργάζεται σε νυχτερινές ώρες ή ε, θέλει να κάνει, υπερορι... κάνει υπερορίες θα πρέπει να μπορεί εφόσον δεν θέλει να απόσχει. Εάν όμως θέλει να διατηρήσει αυτή τη δυνατότητα δεν μπορούμε εμείς να τις επιβάλλουμε να μην το κάνει. Εάν θεωρεί ότι μπορεί ας το κάνει. Θα πρέπει να έχει την ελευθερία επιλογής δηλαδή η γυναίκα. Τώρα για το, χρηματοπιστω... το πλαίσιο της χρηματοπιστωτικής, της οικονομικής κρίσης την οποία διανύουμε. Ε, σαφώς από την πλευρά κάποιων κρατών ε, μελών αυτό δίνει περισσότερα επιχειρήματα για να απορρίψουν τις προσπάθειες βελτίωσης της όλης κατάστασης για το δικό μας θέμα. Όμως εγώ νομίζω ότι ακριβώς σε τέτοιες δύσκολες στιγμές, σε στιγμές δυσχερείς, πρέπει να προστατευτούν ιδιαίτερως οι πλέον ευάλωτοι. Δηλαδή, οι η αλληλεγγύη μας τώρα πρέπει να φαρεί. Και δεδομένων όλων των στόχων που προαναφέραμε για την αύξηση και την καταπολέμηση των δημογραφικών προβλημάτων της Ευρώπης. Ξέρουμε ότι οι Ευρωπαίοι δεν έχουν τόσα παιδιά όσα θα ήθελαν. Αυτό θέλουμε να κάνουμε και εμείς, να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για να τα έχουν οι γυναίκες. Δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να διαλέξουν μεταξύ επαγγελματική σταδιοδρομία και του ρόλου τη μητρότητα. Νομίζω λοιπόν ότι δεν υπάρχουν επιχειρήματα ε, για την χρηματοπιστωτική κρίση, την οικονομική κρίση και τις δυσκολίες που τώρα περνάμε, δεν είναι επιχείρημα αυτό. Επίσης, για τα σημαντικά σίγουρα υπάρχουν κονδύλια από την πλευρά των κρατών μελών. Τώρα, να ευχαριστήσω και το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις τοποθετήσεις τους. Απλώς ήθελα να ξεκαθαρίσουμε το εξής, ότι από την ενιολογική άποψη άλλο πράγμα είναι η γονική άδεια, άλλο η άδεια μητρότητας και άλλο η άδεια πατρότητας. Δεν είναι γονική άδεια ούτε αυτή της μητρότητας ούτε της πατρότητας. Η έννοια που προτείνω εδώ να συμπεριληφθεί και αυτή η διεύρυνση του όλου πεδίου που προτείνω είναι καθοριστική. Η άδεια πατρότητας είναι σημαντική να αναλάβουν και οι πατεράδες και οι μητέρες τη ευθύνη τους. Για την ανατροφή των παιδιών και από τη στιγμή του τοκετού αμέσως πρέπει να αναγνωριστούν στον άνδρα, στον πατέρα τα δικαιώματα αυτά. Γιατί να μην έχει ο πατέρα το δικαίωμα να μείνει, να κρατάει το μωρό του τους πρώτους μήνες της ζωής τους. Το Σαββατοκύριακο συγκεκριμένα στην Πορτογαλία παρέστην σε δημόσια κρόαση για το θέμα αυτό. Μαζί με τον Υπουργό Εργασίας και Αλληλεγγύης της χώρας μας. Και έλεγε ο ίδιος ότι όταν, ήταν πατέρας πρώτη φορά, όταν έγινε πατέρας πρώτη φορά χρειάστηκε να απουσιάσει από τη δουλειά του για να μείνει κοντά στην κόρη του. Και αυτό 20 χρόνια και πριν. Τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ εντωμεταξύ. Οι ανάγκες, η αντίληψη των ευθυνών των ίδιων των πατεράδων από, την, από τη δική τους την πλευρά είναι, έχει αλλάξει, είναι πιο συνειδητοποιημένη. Αυτό λοιπόν για, την, για το καλό του παιδιού, για το καλό των πατεράδων, για να μπορέσει, να μπορέσει να υπάρξει ο συνδυασμό επαγγελματικού και οικογενειακού καθώ και ιδιωτικού βίου τόσο για άντρε όσο και για γυναίκε, απαιτεί αυτή τη στιγμή στο πλαίσιο αυτή τη οδηγία να προβλέψουμε την έννοια τη άδεια πατρότητα. Είναι ένα δικαίωμα που πρέπει να διαθέτει ο κάθε πατέρα και το κάθε παιδί. Η συναισθηματική δεσμή δεν είναι πιο σημαντική για τη σχέση μητέρας-παιδιού από ότι πατέρα-παιδιού και υπάρχουν και καταστάσεις όπου χρειάζεται η παρουσία του πατέρα και πολλές φορές δημιουργείται και καλύτερη συναισθηματική διασύνδεση με τον πατέρα από ότι με τη μητέρα. Εφόσον μάλιστα ο πατέρα ήταν περισσότερο παρόν κατά του πρώτου μήνε τη ζωή του παιδιού από ότι η μητέρα. Εξού λοιπόν και αυτή η διεύρυνση που ζητούμε και για την προστασία της υγείας, της καλής υγείας και της ευμερίας των παιδιών και της μητέρας. Και το λένε και οι ιατρικές μελέτες. Το λένε οι επιστήμονες ότι έξι εβδομάδες μετά τον τοκετό είναι σαφώς υποχρεωτικές, ούτως ή άλλως για να μπορέσει να ανακτήσει την ε, κατάσταση του οργανισμού της η γυναίκα. Εγώ ευτυχώ θα προτείνω ούτω ή άλλω 20 εβδομάδε για την μητέρα, αλλά δύο επιχρεωτικέ εβδομάδε για τον πατέρα και δύο προαιρετικέ. Νομίζω ότι αυτή είναι μια συμβολή που μπορούμε να δώσουμε στην κοινωνία μα για να ξεπεράσουμε συγκεκριμένε προκαταλήψει και να καταπολεμήσουμε και κάποια στερεότυπα. Στερεότυπα που εμένουν. Ο χρόνος αυτό που μπορεί να περάσει κανεί με το παιδί του στου πρώτου μήνε τη ζωή του είναι να αναφέρει το δικαίωμα κάθε γυναίκα αλλά και κάθε άνδρα. Γι' αυτό θέλουμε αυτέ τι αλλαγέ στο σύγχρονο βίο να τι αντικατοπτρίσουμε και στη δική μα την οδηγία και τι προτάσει μα. Με νέε έννοιε, με νέε ανάγκε που έχουν προκύψει. Σήμερα είναι υπαρκτά όλα αυτά στην κοινωνία μα. Θέλω λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε ότι άλλο πράγμα είναι η γονική άδεια, θα το δούμε στο πλαίσιο άλλη οδηγία, άλλο η άδεια μητρότητα και άλλο η άδεια πατρότητα. Η μητρότητα και η πατρότητα είναι δικαιώματα θεμελιώδη και πρέπει να τα δούμε από κοινού και με τρόπο διαρθρωμένο και αλληλοσυμπληρωματικά. Με όλε λοιπόν αυτέ τι συνεισφορέ και τι συμβολέ σα υπόψη, θα συνεχίσουμε να βελτιώνουμε και να επεξεργαζόμαστε αυτή την πρόταση οδηγία. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, εμείς ευχαριστούμε για την δευτερολογία και τα συμπράσματά σα. και πρέπει να σας πω ότι η συζήτηση της εκθέσεως θα γίνει κατά την έκτακτη συνεδρίασή μας στο Στρασβούργο στις 9 Μαρτίου. Τώρα, το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η συζήτηση μιας εκθέσεως. Αφορά την ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στο πλαίσιο των εργασιών των επιτροπών και αντιπροσωπιών. Η συγγέντρια είναι η υποφαινόμενη. mainstreaming για τις εργασίες επιτροπών και αντιπροσωπιών. Πρόκειται για την δεύτερη κατά σειρά έκθεση την οποία έχουμε συντάξει, η πρώτη δε, έγινε το 2006. Θέλουμε να εφαρμόσουμε το ψήφισμα του 2003 όσον αφορά την, ε, το, το mainstream της ε, ισότητας των φίλων στις εργασίες του Κοινοβουλίου. Σαν αρχή λέγαμε θα πρέπει να συνδέσουμε μια τέτοια κρίση σε τέτοια βάση ε, και στη συνέχεια βέβαια κρίθηκε ότι δύο φορές σε κάθε κοινωνική θητεία θα γίνεται μια τέτοια έκθεση. Τάτο σπράβα μπορεί Όσον αφορά τώρα το κείμενο, πρέπει να σας πω ότι στηρίχθηκα στις απαντήσεις ενός ερωτηματολογίου που διανεμήθη σε όλους σε όλες τις επιτροπές, σε όλες τις αντιπροσωπείες. Εκεί κάποιος ε, συνήθως αντιπρόεδρος ή πρόεδρος μάζεψε τις απαντήσεις. Αυτός θεωρείται ο υπεύθυνος για το mainstreaming. Όλες δε οι επιτροπές και οι 21 έλαβαν το αριθμοτολόγιο, 19 απάντησαν εγκαίρως μία απάντησε καθυστερημένο μετά τη λήξη της προθεσμίας και μία δε ε, επιτροπή δεν απάντησε καθόλου Έχετε πάντως λάβει τα αποτελέσματα σε παράρτημα οπότε και μπορείτε να δείτε ε, πώς αναλύονται αυτές οι απαντήσεις πάντως και εγώ τρομπώ να σας πω κάποιες παρατηρήσει δικές μου θεωρούν είναι σημαντικές πρώτα πρώτα να δούμε τι ισχύει και με τη δική μας επιρροή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί είναι αυτό το θέμα το οποίο συνδέεται πάρα πολύ στενά με την εκθέση αυτή γιατί θέλουμε όλες οι επιτροπές και όλες οι αντιπροσωπείες να εργάζονται λαμβάνοντας υπόψη την ισότητα των φίλων. Είχαμε πει να υπάρχουν κάποιοι ε, αρμόδιοι υπεύθυνοι σχετικά με αυτό. Όμως το ότι πίσω υπάρχουν και κάποιες ε, τάσεις να μεταβληθεί το καθεστώς που διέπει την Επιτροπή μας. και να έχουμε ρόλο περισσότερο συμβουλευτικό. Επίσης υπάρχει και μια άλλη τάση σύμφωνα με την οποία θα πρέπει η Επιτροπή μας να διέπεται ακριβώ από όσα διέπουν τις άλλες επιτροπές. Ε, οι συντονιστές διαπίστωσαν ότι αυτό μπορεί να αποτελεί κίνδυνο να υποβαθμίσει ε, τη θέση μας και ε, γι' αυτό και είπαμε επανειλημμένα ότι θα πρέπει ε, να συνεχίσουν να ισχύουν όσα ισχύουν και σήμερα στην Επιτροπή μας. Πάντως, διαπιστώνουμε κάποια βελτίωση στην υπόθεση αυτή. Ε, δηλαδή, η διάρθρωση του προσωπικού στο Κοινοβούλιο από το 1979, το 1979 έχει διπλασιαστεί ο αριθμός των ευρωβουλευτών γυναικών. Ο, όμως θεωρούμε ότι αυτό το 30% που είναι το ποσοστό των γυναικών βουλευτών στο Κοινοβούλιο δεν είναι αρκετός ικανός αριθμός και επίσης θα πρέπει να δούμε τι γίνεται στην διοίκηση του Κοινοβουλίου, τι γίνεται στις γενικές διευθύνσεις όπου η αναλογία είναι δυσμενέστερη. Ε, εκεί δεν έχουμε ούτε το 10%. Η δική μου έκθεση αυτό που θέλω να προβάλλω είναι το εξής. Οι γραμματείες θα πρέπει να ενισχυθούν. Θα πρέπει να έχουν περισσότερη οικονομική υποστήριξη αλλά και περισσότερο προσωπικό ούτως ώστε έτσι να είναι πιο εύκολο ε, το να προωθήσουμε το στόχο μας της ισότητος. Επίσης Κάτι άλλο το οποίο λέω στην εκθεσή μου είναι ότι το κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι υπόδειγμα. Θα πρέπει να είναι παράδειγμα προς για τα εθνικά κοινοβούλια που και αυτά θα πρέπει να διαποτεπώζονται την αρχή της ισότητας των φύλων. Άρα θα πρέπει να αναδεικνύουμε τις άρσεις των πρακτικών Ε, αλλά και να κοιτάμε να εφαρμόζονται αυτές οι αρχές, οι πρακτικές σε εθνικό επίπεδο. Ευχαριστώ την κυρία Κράτσα, την πρόεδρο της ε, ομάδας εργασίας της. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμη αυτή η Επιτροπή για τη δουλειά που κάνει για να συνδέσει την εξωτερική πολιτική με την, εξωτερική, εσωτερική πολιτική του Κοινοβουλίου. Αυτά για την ομάδα αυτή υψηλού επίπεδου. Τώρα δεν θέλω ε, να μακρηγορήσω γιατί όπως σας προείπα στην εκθέσή μου έχω μία ανάλυση ενδελεχή των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου. Εκεί μπορείτε να δείτε τι γίνεται, τι κάνουν οι επιτροπές για το mainstreaming. Ε, κάποιες επιτροπές, ε, όπως θα δείτε, έχουν ένα σχεδίο δράσης. Η Περιφερειακή Επιτροπή, η Επιτροπή Άμυνας, η ε, Επιτροπή Αλληλείας και στις απαντήσεις τους έχουν και κάποιες προτάσεις, προτάσεις για να βελτιωθεί η κατάσταση στο μέλλον. Πάντως θέλω επίσης να ευχαριστήσω τη γραμματεία μας, διότι παρά κάποια σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν όσον αφορά του προσωπικού ανθρώπινου πόρους, ε, χειρίστηκε σε προτεραιότητα αυτή την ε, έκθεση που δεν ήταν εύκολη γιατί υπήρχαν ε, δυσκολίες όσον αφορά την εξεργασία των αποτελεσμάτων. Οπότε, με την ευκαιρία που μου δίνετε τώρα, ευχαριστώ τη γραμματεία μας για όλες τις προσπάθειες. Ευχαριστώ και εσάς που με ακούσατε και τώρα μπορούμε να συζητήσουμε την έκθεση. Α, και κάτι άλλο, μια τελευταία παρατήρηση. Καλέσαμε τους επικεφαλής των αντιπροσωπιών, τους αντιπροέδρους, ε, όλους όσους ασχολούνται με την ισότητα των φύλων να έρθουν στη σημερινή μας συνεδρίαση. Δυστυχώς βέβαια υπάρχουν και άλλες συνεδρίες που γίνονται ταυτόχρονα. Έχουμε πάντως εκπρόσωπο ε, της αντιπροσωπείας για τον Κάφκασο ε, ήρθε, αν δεν ήρθανε, απασχολημένοι. Οπότε τώρα θα δώσω στον συνάδελφο το λόγο. Ah, euh, Α, πρώτα πρώτα κυρία Κράτζα. Πρώτα κυρία Κράτζα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο και σας ευχαριστώ πολύ για την ε, παρουσίαση αυτής της εργασίας που μας κάνατε. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή τη στιγμή και ε, πρέπει να, την, ε, της αποδώσουμε πραγματικά τη σημασία που έχει για την αξιοποίηση του έργου της Επιτροπής μας, για την επίτευξη των στόχων της ισότητας και της ένταξης της διάστασης του φύλου σε όλη την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης σαν ένα αποτέλεσμα της εργασίας που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια γιατί ε, οδεύουμε προς το τέλος της κοινοβουλευτικής ε, περίοδου και όλοι έχουμε έννοια για τον απολογισμό μας και σε αυτά που θα αφήσουμε ε, σαν βάσεις για, την επόμενη, <clears throat> για το επόμενο κοινοβούλιο. ήθελα να, να σταθώ κυρία Πρόεδρε στο γεγονός ότι η, η, η έκθεση αυτή που μας παρουσιάσατε έχει να κάνει, επιτρέψτε να κάνω και εγώ μια μικρή, μια παρουσίαση του στόχου για τα μέλη τα οποία δεν έχουν παρακολουθήσει ε, παλαιότερα, έχουν και καινούργια μέλη στην Επιτροπή μας παλαιότερα αυτό το στόχο. Η, η, πολιτική ισότητα είναι άμεσα συνδεδεμένη με, με την ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές. Έχει μια ιδιαιτερότητα λοιπόν η πολιτική που παράγουμε εδώ, Πώ θα μπει στις πολιτικές των άλλων κοινοβουλευτικών επιτροπών, των άλλων πολιτικών εκφράσεων του Κοινοβουλίου. Ε, και αυτό συνδέεται με τη δημιουργία του High Level Group που προσπαθεί να αξιοποιήσει τη δουλειά που γίνεται εδώ και να την ε, ε, διοχετεύσει στις άλλες επιτροπές. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, επειδή όπως ανέφερε και κυρία Πρόεδρος, έχω την τιμή να μοναθέσει ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου την Προεδρία αυτού του high Level Group, έχουμε συνεργαστεί με την Επιτροπή Γυναικών και με την κυρία Ζαμπόσκα προσωπικά που είναι μέλος αυτού του High Level Group, πώς θα επιτευχθεί η αξιοποίηση της δουλειάς που γίνεται εδώ μέσα στις άλλες εργασίες του Κοινοβουλίου. Πρώτον, στις κοινοβουλευτικές επιτροπές το, το, το ερωτηματολόγιο που παρουσίασε η κυρία Ζαμπόσκα δείχνει ότι δεν έχει συνειδητοποιηθεί αυτή η ανάγκη. Ούτε τα κατάλληλα μέσα έχουν διατεθεί στις γραμματείες των επιτροπών, η γραμματεία η δική μας η οποία κάνει ένα αξιόλογο έργο και δίνει τη βοήθειά της και τις συμβουλές στις άλλες επιτροπές, χρειάζεται πολύ περισσότερο προσωπικό και υλικέ δυνάμει για να μπορέσει να αντιμετωπίσει όλε αυτές τις ανάγκες. Άρα πρώτον πρέπει να τονίσουμε την ανάγκη να ενισχυθούν με ανθρώπινο δυναμικό και με εκπαίδευση οι γραμματείε των άλλων επιτροπών. Δεύτερον, να λειτουργήσει το σύστημα των συνδέσμων μας, όπως είναι ο συνάδελφος από την αντιπροσωπεία στον Κάφκασο που θα, που θα μιλήσει σε λίγο, των συνδέσμων στις άλλες επιτροπές. Υπάρχει μια ήδη επιτροπή που ανέφερε ο κ. Ζαμπόσκο που δεν έχει καν απαντήσει στο ερωτηματολόγιο. Σημαίνει ότι δεν έχει ληφθεί σοβαρά υπόψη αυτή η υποχρέωση που ανέλαβαν οι κοινοβουλευτικέ επιτροπέ. Θεωρώ πολύ σημαντικό και πιστεύω ότι το συμμερίζεστε ότι με τη δική μου πρόταση στο High Level Group επεξετάθη η ανάγκη αυτή και στις αντιπροσωπείες. Διότι η Επιτροπή μας έχει πολλές φορές τονίσει τη σημασία που έχει η διάσταση του φύλου στην ανθρωπιστική στην αναπτυξιακή στην πολιτική μας σχέση με, ε, γενικά στις εξωτερικές σχέσεις ένωσης. άρα λοιπόν το λέω αυτό με έμφαση κυρία πρόεδρε επειδή τυχαίνει να είμαστε όλες εδώ μέλη άλλων επιτροπών να έχουμε την έννοια της παρακολούθησης και εμείς πως αυτό λειτουργεί στις άλλες επιτροπές. επίσης θέλω να τονίσω κάτι το οποίο το είπατε, επιτρέψτε μου να το ξαναπώ κι εγώ, ότι η προσπάθεια αυτή αξιοποίησης της δουλειάς, του ρόλου της Επιτροπής Γυναικών, της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές του Κοινοβουλίου, δεν έχει να κάνει με αλλαγή του ρόλου και της θέσης της Επιτροπής Γυναικών. Πρέπει στην αναθεώρηση του Κοινοβουλίου να στηρίξουμε τα δικαιώματα, την αναβάθμιση και όχι την υποβάθμιση της Επιτροπής αλλά λόγω της ιδιαιτερότητας αυτής της επιτροπής πρέπει η εργασία μας να γίνεται και στις άλλες επιτροπές. Ε, αυτό ήθελα να τονίσω κυρία Πρόεδρε και ε, πιστεύω ότι εμείς που είμαστε, πολλές είμαστε σταθερά μέλη αυτής της Επιτροπής χαίρομαι που νέοι συνάδελφοι που έρχονται ή με τη διεύρυνση ή αν καθιστώντες άλλους συναδέλφους εντάσσονται σε αυτή την Επιτροπή. Είναι μια καλή ευκαιρία λοιπόν όλοι μαζί να πετύχουμε τους στόχους της αναβάθμισης της Επιτροπής μας αλλά και της διοχέτευσής της και της επιρροής της στις άλλες πολιτικές του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ πολύ και για την παρουσία και για τη συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κράτσα. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχετε το λόγο εσείς τώρα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, πρώτα-πρώτα που μας ε, προσκαλέσατε τις επιτροπές και τις ε, αντιπροσωπείες. Αρμενία, Γεωργία και Αζερμπαϊτζάν είναι τα δικά μας θέματα και ανταποκριθούμε στην επίσκεψή σας ε, για την οποία προετοιμαστήκαμε σύντομα σε συνεργασία με την κυρία Σλερ Μπεγγέν και όσον αφορά τη δική μας δουλειά. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε κάνει και τρομερά πράγματα και δεν το λέω τόσο αρνητικά. Θα σε εξηγήσω τι εννοώ. Το βασικό θέμα για τις αντιπροσωπείες είναι πώς θα εντάξουμε στις εργασίες μας αυτό το gender mainstream, την ισότητα των γυναικών, πώς αυτό θα εφαρμοστεί στις αποστολές, ε, στα όργανα της αντιπροσωπείας μας, σε όλη τη δουλειά. Γιατί όντως καταβάλαμε μια προσπάθεια για τέτοια ζητήματα, για ανθρώπινα δικαιώματα, για κάθε ε, προσπάθειά μας, κάθε πρωτοβουλία μας. διαπίστωση τώρα είναι ότι προσπαθούμε σε κάθε, μας προσπάθησε σε κάθε ενέργεια να περάσει και το μήνυμα της ισότητας ανδρών και γυναικών. Στέκομαι τώρα σε αυτό το, το θέμα της έκθεσης, το ότι η κάθε αντιπροσωπεία και επιτροπή για την ισότητα των γυναικών έχει τη δική της άποψη για την καθημερινή της δικές της ιδιορυθμίας. Όσον τώρα τα δικά μας θέματα, τον Κάφκασο κλπ. Σε συνεργασία με την κυρία Ζελεμπανιά καταλήξαμε στο ότι οι χώρες αυτές με τις οποίες ασχολούμεθα για ιστορικούς λόγους, τον 20ο αιώνα ασχολήθηκαν με την ισότητα των φίλων κάτι το οποίο ισχύει βέβαια για κάθε κοινωνία, για όλο τον κόσμο. Και πολλές φορές αναδεικνύει το θέμα αυτό στις επαφές μας με τις χώρες αυτές. Πέρσι, όπως ξέρουμε, είχαμε και τον πόλεμο στον Κάφκασο, και στα πλαίσια του πολέμου αλλά και κάθε άλλη κρίση που σοβεί ή που υφέρεται συζητήσαμε και αυτό το θέμα όπως και άλλα κλαδικά, οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και όπως προείπα δεν έχουμε κάνει καμία εντυπωσιακή σαν πρόοδο, όμως διαπιστώνεται ότι οι ομόλογοι μας από τις χώρες εκείνες πολλές φορές έχουν πολύ περισσότερες γυναίκες σύνδεσή τους από τη σύνθεση των δικών μας αντιπροσωπιών που πάνε εκεί για μια αποστολή. Να, κάτι θετικό. θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε λέγοντας ότι κάνουμε μια αφετηρία από τώρα, έχουμε την, το, το έργο αυτής της ομάδας υψηλού επίπεδου, οπότε και θα προχωρήσουμε ούτως ώστε σταθερά και μόνιμα και συνέχεια το mainstreaming να το λαμβάνουμε υπόψη σε όλη μας εργασίες. Να μην θεωρείται ένα πρόβλημα σημειακό, αλλά να υπάρχει μια συνέχεια, να είναι χαρακτηριστικό πάγιο όλων των δραστηριοτήτων μας. Ε, Η πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Ε, κύριε Γκόμες έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα για την έκθεση που έχουμε στα χέρια μας Σε ό,τι αφορά τον τρόπο που αντιμετωπίζει τα ζητήματα των δύο φίλων η Επιτροπή αυτή και από αυτή τη σκοπιά, είναι πολύ σημαντικό το έργο που έχει γίνει, αλλά ακόμη απέχουμε πολύ από το να καλύψουμε όλες τις ανάγκες που υπάρχουν. Όπως, όπως προείπε ο συνάδελφος, ο τομέας αυτός, ένας τομέας όπου εμπλέκονται οι γυναίκες και εξορισμού αφορά τις γυναίκες, γιατί πολλές φορές οι πρόσφυγες, όπως γνωρίζουμε, είναι γυναίκες και παιδιά. Και βλέπουμε σήμερα όλο και περισσότερο οι συγκρούσεις, οι σύγχρονες ε, σειράξεις να αφορούν άμεσα τις γυναίκες και ως στόχους προεπιλεγμένους και να είναι στόχος ακριβώς των, ενός πολέμου. Ενώ λοιπόν υπήρξε συνειδητοποίηση του θέματος αυτού από τις δομές και τους σχηματισμούς του Συμβουλίου της Επιτροπής και του δικού μας του Κοινοβουλίου για την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι δικές ανάγκες των γυναικών από την άποψη της άμυνας και της ασφάλειας και ιδίως να εξασφαλίσουμε τα δικαιώματα των γυναικών αυτών που θα μπορούσαν να είναι και ενεργοί προαγωγή, προ, προωθητές των, ε, της άμυνας και της ασφάλειας, παρόλα αυτά βλέπουμε ότι ο δρόμος που πρέπει ακόμα να διανύσουμε είναι μακρύς. Υπάρχουν ε, ούτω ή άλλω σε αποφάσει τα ψηφίσματα 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, παλιότερα ψηφίσματα που επιβάλλουν την ε, επιπλέον την περαιτέρω συμμετοχή και εμπλοκή των γυναικών στην ειρήνευση και την πάυση ανθρωπραξιών γενικώ και ένα άλλο ψήφισμα το πρόσφατο, φετινό και πάλι του Συμβουλίου Ασφαλείας το 1820 το οποίο ακριβώς χαρακτηρίζει ως εγκλήματα πολέμου τα εγκλήματα κατά των γυναικών, ε, βιασμούς, εγκλήματα σεξουαλικού χαρακτήρα και ούτω Πράγματα που βλέπουμε να συμβαίνουν συνεχώς βεβαίως στις σύγχρονες εμπόλεμες συγκρούσεις. Έχουμε δει τι προβλήματα υπάρχουν σχετικά. Έχουμε δει τις αποστολές της ΠΕΖΔ, της κοινή ασφάλειας, της κοινή πολιτικής άμυνας και ασφάλειας. Είδαμε το τι συνέβη στην αποστολή στο Κονγκό το 2006, την αποστολή στη Γουινέα Μπισάου Μια αποστολή που πρέπει να ασχοληθεί με τη μεταρρύθμιση του τομέα άμυνας και ασφάλειας της χώρας αυτής. Και εκεί υπήρξαν προβλήματα, προβλήματα ακριβώς με τα δικαιώματα των γυναικών. Ακόμη δεν έχουμε μορφυλοποίηση όλων αυτών των ψηφισμάτων. Από την πλευρά του Κοινοβουλίου και όπως και σε πολλά σημεία αναφέρεται εδώ στην έκθεση σημαντικός είναι ο ρόλος κάποιων επιτροπών όπως τους 11 και λέγεται ότι 21% των ε, μελών που συμμετέχουν είναι γυναίκες. Αυτό όμως έχει μια επιπλέον σημασία. Διότι τρεις από τους συντονιστές των διαφορών επιτροπών είναι γυναίκες των ε, σοσιαλιστών εγώ ίδια, των φιλελευθέρων και των πρασίνων επίσης. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι γυναίκες επηρεάζουν την εργασία του κοινοβουλίου αυτού. Και άλλωστε, στο πλαίσιο αυτής της Επιτροπής, ας δούμε και κάτι παραπάνω. Ότι υπάρχει και μια επιπλέον στήριξη για γυναίκες από διάφορες χώρες, όπως αυτές του κοσφοπεδίου. Εκεί διευκολύναμε και την εργασία της αποστολής Γιούλεξ στο Κωσυφοπέδιο, όπως θυμάστε. Και πρόσφατα είχαμε και μια αποστολή της ΕΝΤΕ στο Κωσυφοπέδιο. Συζητήσαμε με τις γυναίκες αυτές και οι γυναίκες αυτές μας λένε ότι για την ώρα έχουν ακόμη κάποιες δυσκολίες, αρκετές δυσκολίες. Γιατί παρά την αποστολή Γιούλεξ, παρά το εστιακό το σημείο επαφής που έχει δημιουργηθεί για συντονισμό με τους υπευθύνους των αποστολών αυτών, τελικά ε, έχουν ακόμα προβλήματα και είναι εκείνες που έκαναν έκκληση προς το Κοινοβούλιο για να ασχοληθούν με τα ζητήματα ισότητας των δύο φίλων στη χώρα τους. Είναι ζητήματα που ζήτησαν να περιληφθούν στη δική μας την πολιτική ατζέντα. Άρα εδώ μας ενδιαφέρει όχι μόνο τις διαφορές μπορεί να κάνει, να έχει η συμμετοχή των γυναικών σε τέτοιου είδους ε, ένοπλες σειράξεις, αλλά και πώς ενεργά μπορούν να συμμετέχουν οι γυναίκες για τους αντίθετους στόχους από αυτούς των πολέμων. Θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε και ως Επιτροπή να επαγρυπνούμε για τα θέματα αυτά. Γιατί είναι ο πιο ζωτικός ρόλος που μπορούμε να έχουμε σε αυτά τα θέματα. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κυρία Γκόμες. Μας μένουν περίπου 10 λεπτά. Είναι πολλοί οι συνάδελφοι που ζητούν το λόγο, αλλά θα πρέπει να προσπαθήσετε να συντομεύσετε, γιατί στη συνέχεια έχουμε και τη δημόσια ακρόαση. Κυρία Πλεστίνσκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι η έκθεση συνολικά είναι καλή. Δεν μπορούμε παρά να χειροτήσουμε τη δουλειά σας. Είναι πολύ καλή προσέγγιση σας. Είναι πολύ σημαντικό ότι βασιστήκαμε εδώ και σε ερωτηματολόγια. Κάτι όμως που μπορεί κανείς να αναρωτηθεί είναι πόσο σοβαρά έλαβαν υπόψη οι επιμέρους επιτροπές στο εν λόγω ερωτηματολόγιο. Και για τη συζήτηση του όλου θέματος ε, όχι μόνο να συζητήσουμε θεωρητικά το θέμα είναι ενδιαφέρον, αλλά πώς πρακτικά στην καθημερινή ζωή υλοποιούνται οι σχετικές διατάξεις. Ε, γιατί εμείς λαμβάνουμε αποφάσεις, προτείνουμε μέτρα, αλλά πολλές φορές οι άλλες επιτροπές παραβλέπουν όλα αυτά και όχι μόνο το 100%, δεν ότι δεν υλοποιούν το 100%, αλλά το 10% κάποιες φορές δεν λαμβάνουν υπόψη. Από την πείρα μας είδαμε ότι όταν οι συστάσεις δεν εφαρμόζονται στην πράξη γενικώ, χρειάζονται κυρώσει. Ε, λόγου χάρη η εσωτερική αγορά δεν θα μπορούσε να έχει δημιουργηθεί αν δεν επιβάλλονταν και κυρώσει. Δεν ξέρω εδώ τι κυρώσει θα έπρεπε να επιβάλλονται, διοντολογικέ, ηθικέ, οικονομικέ, ε, ακόμη και στο Ευρωκοινοβούλιο. Δεν ξέρω πώ θα μπορούσαν οι επιτροπέ να αναλάβουν περισσότερε ευθύνε από το θέμα, να ευαισθητοποιηθούν ω προ αυτό. Πρόεδρο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πλουσίνσκα. Επισημάνατε νομίζω με πολύ μεγάλη ακρίβεια τα προβλήματα. Η κυρία Πρέτση έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε μία επισκόπηση της ε, επιρροής που μπορεί να έχει η Επιτροπή των Γυναικών και στις άλλες επιτροπές, ιδιαίτερα τώρα πριν από τις εκλογές και ιδιαίτερα εν ώψη της νέας θητείας που θα ξεκινήσει, για να είμαστε θέση να αποδείξουμε ότι χρειάζεται να ληφθούν νέα μέτρα στην νέα θητεία. Περισσότερες γυναίκες πρέπει να αναλάβουν ηγετικές θέσεις στις, ε, στα όργανα του Κοινοβουλίου. Περισσότερες γυναίκες πρέπει να είναι πρόεδροι στις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Αυτό είναι σημαντικό. Το διεκδικούμε εδώ και χρόνια βέβαια. Επί τη βάση όμως της εκθέσεως αυτής, επί τη βάση των τελευταίων τοποθετήσεων και επιχειρημάτων που μπορούμε να προβάλλουμε, έχουμε περισσότερο, ε, περισσότερο επιθό, θα έλεγα. Βεβαίως θα δούμε πώς θα αντιμετωπίσουν το ζήτημα αυτό και τις προτάσεις μας οι άντρες, αλλά πρέπει και εμείς οι γυναίκες να ενωθούμε, να αγωνιστούμε μαζί. Πολλές φορές έρχονται εκθέσεις και δεν κερδίζουμε παρά την παρουσία αρκετών γυναικών μέσα στις, ομάδες, στις επιτροπές μας. Είχαμε συμφωνήσει παραδείγματι την ανάθεση των θεμάτων αυτών σε μια εκπρόσωπο των γυναικών για τα θέματα της γυναίκας, διαμεσολαβητή θα έλεγα. Πώς τα θέματα αυτά τα χειρίζεται, πώς στην πράξη αντιμετωπίζονται τα προβλήματα και νομίζω ότι με αυτό με αυτή τη δυνατότητα, με αυτούς τους υπευθύνους ανθρώπους μπορούμε να έχουμε μέσα σε επιτροπές, μπορούμε να βρούμε τις λύσεις. Πολλά μένουν ακόμη να γίνουν, αλλά νομίζω ότι αν όλοι μαζί καθίσουμε καλά και επεξεργαστούμε μια νέα στρατηγική για την προσεχή θητεία, θα κερδίσουμε πολλά. Και επίσης, σε θέματα που έχουν να κάνουν με την ε, έγκριση την αποδοχή καλύτερα των εκθέσεων μας από τις άλλες επιτροπές. Βλέπουμε δυστυχώς ότι ε, συχνά ε, διαγράφονται οι δικές μας τροπολογίες, δεν, δεν περνούν όπως θα, θέλανε, όπως θα θέλαμε από τις υπόλοιπες επιτροπές. Εγώ θα ήθελα ο συντονίστρια κιόλα να κάνω μια καλύτερη προσπάθεια. Ξέρω ότι δεν είμαστε αρκετά αποτελεσματικέ στι προσπάθειέ μα αυτέ. Και αν κοιτάξουμε και τι στατιστικέ από τι 18 επιτροπέ που αξιολογούνται εδώ μέσα, οι 7 έχουν ποσοστό κάτω του 30% σε επίπεδο αποδοχής των προτάσεών μας και αυτό πραγματικά είναι λόγος ανησυχίας. Ας ενισχύσουμε λοιπόν τις προσπάθειές μας και ας προβάλλουμε τα, τις θέσεις ε, που ακούστηκαν εδώ και μάλιστα πριν από την εκκίνηση της νέας θητείας. Η Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρέτση. Κυρία Μικέλης Ράμος έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα ζητώ να με συγχωρήσετε που άργησα να έρθω αλλά τα πράγματα είναι πολύ ζόρικα για μένα αυτή τη βδομάδα. Πάντως θέλω να σας αναφέρω ότι θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή αυτή η έκθεση, είναι πάρα πολύ καλή αφετηρία, ούτω ώστε το Κοινοβούλιο να ασχοληθεί ουσιαστικά με αυτό το θέμα. Εγώ εδώ είμαι την πρόεδρος και διεκπροσωπώ την Επιτροπή της Αλληλείας για να δούμε πώς θα εντάξουμε στις δουλειές μας, στις εργασίες μας, την υπόθεση της ισότητας, ό,τι πρωτοφορές ζητήσατε σας τη στείλαμε και πρέπει να σας αναφέρω ότι ως επιτοπλίστων οφείλεται αυτό στην ευαισθησία του ε, ε, συναδέλφου, τη συναδέλφου της κυρίας Κρέσπο που είναι υπεύθυνη της γραμματείας μας για αυτά τα θέματα είναι εδώ στην αίθουσα μαζί μας επίσης μην ξεχάσω να σας πω ότι το είπαμε και στις απαντήσεις μας το ότι Υπάρχει ένα μεγάλο κενό γνώσης πληροφορίας όσον αφορά τα γυναικεία θέματα σε σχέση με την αλία. Αυτό το κενό προσπαθούμε να το άρουμε ε, και έτσι να δουλέψουμε πιο καλά στην επόμενη κοινοβουλευτική θητεία. Επίσης, θέλω να σας πω ότι ντρέπομαι. Ντρέπομαι γιατί έχουμε τόσο χαμηλή συμμετοχή των γυναικών στην Επιτροπή μας. 22,2% μόλις. Πάντως, από την άλλη μεριά, ε, κάποιες από αυτές τις γυναίκες συμμετέχουν στο Προεδρείο. Τρεις συντονίστρες έχουμε, αλλά και τρεις αντιπροέδρους. Οπότε, ε; κάπως εξισορροπούνται τα πράγματα. Όπως και να είναι, θέλαμε ε, όσο γίνεται περισσότερο να εκπροσωπούνται οι γυναίκες στις εργασίες μας και συγχαρητήρια Πρόεδρε για την ε, πάρα πολύ αξιόλογη εκθεσή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ ιδιαίτερως και την Επιτροπή που κάλεσε την Χάριετ Χάρμαν να μας μιλήσει σήμερα το απόγευμα. Όπως γνωρίζετε είναι υπουργό μας για θέματα γυναικών του Ιωμένου Ιδιαίτερα ευχαριστώ την Επιτροπή, την, Πρόεδρο, για την έκθεση αυτή που είναι πάρα πολύ καλή. Είναι βέβαια λυπηρό το ότι δείχνει πόσο κακέ επιδόσει έχει το Ηνωμένο Βασίλειο. Βέβαια και τα άλλα κράτη-μέλη ενδεχομένω, αλλά έχουμε πολύ λίγε γυναίκε εμεί στο Ηνωμένο Βασίλειο στη Βουλή μα. σω λιγότερε από 20% και χειρότερα ποσοστά από ό,τι έχουμε μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει να κάνουμε λοιπόν πολλά για να ενισχύσουμε τη θέση των γυναικών, την παρουσία των γυναικών και μέσα στο Κοινοβούλιο και μέσα στι κοινοβουλευτικέ επιτροπέ. Σα ευχαριστώ ιδιαίτερα για τι προσπάθειέ σα και ιδιαίτερα να υπογραμμίσω τα εξή που υπόθηκαν ήδη. Θα μπορούσε να υπάρχει κάποιος στην Επιτροπή ο οποίος θα παρακολουθεί τα θέματα αυτά των γυναικών και την αποδοχή τους από τις άλλες επιτροπές. Όπως είπατε είναι πολύ καλή ιδέα και πρέπει να τα παρακολουθούμε, να παρακολουθούμε την εξέλιξη των διάφορων θεμάτων γιατί ίσως αποδειχθεί τελικά ότι δεν έχουν τόσο καλή ε, τόσο καλό αντίκτυπο όσο θα θέλαμε. Επίσης θα μπορούσαμε να ε, κάνουμε μια εκστρατεία θα έλεγα ευαισθητοποίηση στις δικές μας τις ομάδες η καθεμία ε, για να πείσουμε περισσότερο να υπάρχουν και πιο πολλές υποψήφιες γυναίκες και, καλύτερες, και καλύτερη θέση για τη γυναίκα, θέσεις συντονιστικές και τα λοιπά μέσα στις ομάδες μας και βέβαια σε επίπεδο Προεδρείου να κοιτάξουμε τι θέσει στην παρουσία των γυναικών, αλλά επίση να κοιτάξουμε και την παρουσία των γυναικών σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί και εκεί, ε, όπω και στο, στα, στα λοιπά θεσμικά όργανα, πάση περιπτώσει η Επιτροπή ιδιαίτερα, πρέπει να δούμε τι παρουσία έχουν οι γυναίκε. Πολλά έχουμε να κάνουμε λοιπόν. Και πρέπει επίση να ξαναδούμε την έκθεση αυτή κάποια στιγμή στο μέλλον για να παρακολουθήσουμε τι αποτελέσματα έφερε. Σα ευχαριστώ πολύ. Λέει Πρόεδρος, κυρία Πέτρα. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και συγχαρητήρια ταυτόχρονα για το έργο σας. Θα ήθελα απλώ να πω δύο λόγια για την αντιπροσωπεία για τη σχέση μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, της οποίας είμαι και εγώ μέλος. Όπως γνωρίζετε έχουμε πρόεδρο γυναίκα στην αντιπροσωπεία αυτή. Καλό λοιπόν αυτό. Βέβαια το θέμα της ισότητας ανδρών και γυναικών είναι διαρκώς παρόν στα θέματα που εξετάζουμε, στη μέρημνα που επιδεικνύουμε. Πριν από δύο εβδομάδες μόλις άλλωστε διεξήχθη μια συνεδρίαση ειδικά αφιερωμένη στα παιδιά που ζουν μόνα τους στη Μολδαβία, ζουν μόνα τους ενδεχομένως γιατί οι γονείς έχουν φύγει στο εξωτερικό για να εργαστούν στις δικές μας χώρες, θα έλεγα. Κατάσταση ιδιαίτερα βέβαια δύσκολη για τα παιδιά αυτά. Και για άλλη μια φορά θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η αντιπροσωπεία μας αυτή για τη σχέσεις της Μολδαβίας ασχολείται με πολύ σοβαρότητα πάντοτε για τα θέματα ισότητας ανδρών και γυναικών. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, σας ευχαριστώ και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που έλαβαν το λόγο στην συζήτηση. Ασφαλώς, ό,τι ε, και να έχουμε επιτύχει μέχρι τώρα χρειάζεται βελτίωση. Πάντοτε χρειάζεται να κάνουμε περισσότερα. Για μια δε ολοκληρωμένη προσέγγιση ως προς την ε, ενσωμάτωση του ζητήματος όταν των δύο φύλων σε όλες τις πολιτικές μας, το mainstreaming που λέμε, πολλά έχουμε να κάνουμε ακόμη μέσα στο κοινοβούλιο. Η δε αναλογία της συμμετοχή των γυναικών στις κοινοβουλευτικέ επιτροπές, νομίζω ότι είναι αρκετά λογική στις περισσότερες από τις επιτροπές μας. Γιατί, Γιατί αν έχουμε βουλευτές γυναίκες κατά 30% εκπροσωπούμενες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τότε και η παρουσία των γυναικών κατά 30% αναλογία μέσα στις κοινοβουλευτικές επιτροπές είναι η σωστή. Δεν μπορούμε να ανατρέψουμε αυτή την αναλογία. Ίσως μάλιστα σε ορισμένες επιτροπές να χαρακτηριστεί αρκετά χαμηλή παρουσία των γυναικών, αλλά υπάρχουν άλλες όπου είναι πολύ έντονη. Άρα περισσότερο θα πρέπει να επιδιώξουμε την εκλογή γυναικών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ένα ζήτημα που υπογράμμισε η κυρία Πλωσίνσκα. Η περιορισμένη αποδοχή των γνωμοδοτήσεών μας από τις άλλες επιτροπές. Όταν εμείς έχουμε λοιπόν γνωμοδότηση ως Επιτροπή των Γυναικών σε κάποια κατουσία, που υποβάλλουμε σε κάποια κατουσία αρμόδια ή καθήλυνα αρμόδια καλύτερα επιτροπή, διαπιστώνουμε μερικές φορές ότι ορισμένες από αυτές τις επιτροπές δεν αποδίδουν την δέουσα σημασία ή τον σεβασμό που θα έπρεπε στη γνωμοδότησή μας ε, παραβιάζοντας ακόμη το άρθρο 47 του κανονισμού. Άρα και μια καλύτερη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής μας και των λοιπόν Επιτροπών χρειάζεται όπως άλλωστε αναφέρθηκε και Ίσως, γιατί θα πρέπει να επισημάνω επίσης ότι από το 2006, από την πρώτη έκθεση αξιολόγησης, ε, είχα ε, την πρωτοβουλία να αναπτύξω επαφές με διάφορους ε, εκπροσώπους επιτροπών άλλων. Δυστυχώς όμως, μόνο δύο ή τρεις θα έλεγα από τους Οι ή αντιπροέδρους των επιτροπών αυτών επέδειξαν ενδιαφέρον για μια τέτοια συνεργασία. Τις περισσότερες φορές δεν προσέρχονταν καν στις συναντήσεις, Έστειλαν βοηθό για να συνομιλήσει μαζί μου και ε, βλέπω ως μειονέκτημα την ανυπαρξία στράτευση από πλευρά των συναδέλφων αυτών. Σε αυτό νομίζω θα πρέπει να επιμείνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ ιδιαίτερα στην κυρία Αντιπρόεδρο και τους ε, προέδρους και αντιπροέδρους των επιτροπών που εκδηλώνουν τέτοιο ενδιαφέρον για τα θέματα αυτά. Για όλους, ευχαριστώ όλους τους αδέλφους που κατέθεσαν ε, προτάσεις και παρατηρήσεις και ελπίζω και η έκθεση αυτή να εγκριθεί στην, ε, από την Ολομέλεια. Προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών έχουμε την 17η Φεβρουαρίου, 12 το μεσημέρι, 17 Φεβρουαρίου, 12 το μεσημέρι, περίπου μια εβδομάδα έχουμε ακόμη δηλαδή στη διάθεσή μας. Η ψηφορία θα γίνει στις 21 Μαρτίου στην Επιτροπή μας. Και προβλέπεται η έγκριση από την Ολομέλεια τον Απρίλιο της εκθέσεως. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια και για τις τροπολογίες βέβαια που θα μπορέσουμε να περιλάβουμε στην έκθεση. Και βέβαια προσμένω να συνεχιστεί η συνεργασία μας αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώνουμε εδώ το ε, τμήμα που αφορούσε τις εργασίες της Επιτροπής μας για το πρωινό μας και ξεκινάμε τώρα την ακρόαση που έχουμε προβλέψει. Κάποια διαδικαστικά. Πρώτα απ' όλα ότι θα διακόψουμε για λίγο για να ανασταθούμε και θα αρχίσουμε σε 2-3 λεπτά. Ευχαριστώ.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 vážené kolegyne συνάδελφοι, ας ε, συνεχίσουμε τώρα με το επόμενο θέμα στην ημερήσια μας διάταξη που είναι η δημόσια κρόαση για το και σε ανωνυμία. ορίζω τους εμπειρογνώμονές μας, τους ειδικούς μας που έχουν έρθει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μας μιλήσουν για να μας μιλήσουν για την εμπειρία τους από την ε, υπόθεση αυτή των τοκετών σε ανωνυμία. Ίσως η επιλογή του θέματος για τη δημόσια κρόαση να εξέπληξε κάποιους εξημών. Πλην όμως πρόκειται για ένα θέμα το οποίο απασχολεί ιδιαίτερα τις γυναίκες. Είναι ένα θέμα διαφιλονικούμενο, συμφωνώ. Είναι ένα θέμα στο οποίο τα κράτη-μέλη δεν έχουν ενιαία αντιμετώπιση ή θέσεις και όμως είναι ένα θέμα στο οποίο πιστεύω ότι πρέπει να συζητήσουμε, διότι έχουμε να κάνουμε ένα νομοθέτημα το οποίο θα πρέπει να προσφέρει στις γυναίκες την επιλογή σε μια κατάσταση δύσκολη, σε μια κατάσταση που με δυσκολία μπορεί να αντιμετωπίσει μια γυναίκα. Όταν δηλαδή ε, διαπιστώσω ότι είναι έγκυος, όταν έρθει η ώρα μετά να γεννήσει, ε, ο θεσμός αυτός του το σε ανωνυμία πιστεύω βοήθησε στο να σωστούν πολλές ε, ζωές παιδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση παιδιών που θα είχαν ε, κινδυνέψει με άμβλωση, ενδεχομένως θα είχαν φωνευθεί αμέσως μετά το τοκετό. Η ίδια προέρχομαι από τη Σλοβακία. Υπάρχει άλλη μια συνάδελφος από τη Σλοβακία εδώ. Στη χώρα μου το θέμα μας έχει απασχολήσει. Το συζητήσαμε το 2004, καθώς ξέσπασε δημόσιο διάλογο όταν βρέθηκε ένα νεογέννητο αγοράκι στο διάδρομο ενό νοσοκομείου και έτσι πολύ γρήγορα αντιδράσαμε για να εισαγάγουμε την νομοθεσία αυτή περί το και σε ανωνυμία. Πρέπει να πω ότι ήταν ακαθόδε το ζήτημα αυτό για τη χώρα μου. Ήταν οδυνηρέ οι συζητήσει. Όχι γιατί κανεί τα τάσσονταν κατά του το και του σε ανωνυμία τόσο, όσο γιατί εκλήθημε να διατυπώσουμε νομοθεσία η οποία θα κάλυπτε και τη στιγμή τη χρονική την περίοδο μάλλον τη χρονική που αφορά τον τοκετό, τη γέννηση του παιδιού, αλλά και τη μετέπειτα περίοδο. Την ενηλικίωση του παιδιού θα προστατεύει το παιδί, θα προστατεύει και τη μητέρα όμως η νομοθεσία αυτή. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με μία σχηματικά θα το πω τριγωνική σχέση, διότι έχουμε να κάνουμε με την δυνατότητα να εξασφαλιστεί η προσφορά αυτού που στην Σλοβακία ονομάζουμε σωτήρια φωλεά, δηλαδή μια κοιτίδα στην οποία μπορεί να αφαιθεί το παιδί, ενώ η μητέρα θα μπορούσε να το γεννήσει στο σπίτι, έρχεται και αφήνει το παιδί στην κοιτίδα αυτή η μητέρα. Η κοιτίδα είναι προστατευμένη με ένα σύστημα συναγερμού που ενημερώνει αμέσως το προσωπικό του νοσοκομείου ότι αφέθηκε ένα νεογνώ ε, στην κοιτίδα αυτή. Υπάρχει λοιπόν η προστασία του νεογνού, υπάρχει δυνατότητα της ε, τούτο και του ανώνυμα μέσα στο νοσοκομείο και βέβαια υπάρχει και το τρίτο σκέλος αυτού του τριγώνου, ολόκληρο το θεσμικό πλαίσιο, οι οργανισμοί, οι φορείς εκείνοι που στηρίζουν την έγκυο γυναίκα όταν έχει ανάγκη. Μπορεί να της προσφέρουν έναν τόπο στον οποίο μπορεί να διαμείνει για να γεννήσει το παιδί της, είτε θέλει επώνυμα είτε ανώνυμα να το γεννήσει, θα της προσφερθεί η μέρημνα και η φροντίδα που χρειάζεται τόσο ίδια όσο και το παιδί της μετά τον τοκετό. Και θεωρώ καλό το ότι το θέμα αυτό μπορέσαμε εμείς στην πατρίδα μου να το καλύψουμε με μια τόσο ευρεία νομοθεσία και να μην περιοριστούμε μόνο στη δυνατότητα να γεννήσει μια γυναίκα το παιδί τη χωρί να δώσει τα στοιχεία τη ταυτότητά τη. Έχουμε λοιπόν πέντε χρόνια εμπειρία από την εφαρμογή τη νομοθεσία αυτή στην ε, Σλοβακία. Τα αποτελέσματα που σημειώνονται είναι καλά και αποτελούν ε, θετική πηγή και βάση για περαιτέρω συζήτηση. Και τώρα επιτρέψτε μου να καλωσορίσω τις πυρογνώμονές μας. Δυστυχώς η τρίτη που θα έπρεπε να έρθει στην συνεδρίασή μας, την οποία είχε προτείνει και η κυρία Μπράιερ και την ευχαριστώ για την πρωτοβουλία της. Διότι με βοήθησε, μας βοήθησε να οργανώσουμε τη συζήτηση γύρω από το θέμα αυτό. Δυστυχώς λοιπόν η κυρία από τη Γερμανία, η εμπειρογνώμων από τη Γαλλία δεν μπόρεσε να προσέλθει στην ακρόασή μας. Ευχαριστώ όμως και καλωσορίζω τις δύο εμπειρογνώμονες, την κυρία από την Ελλάδα και την ε, άλλη κυρία από τη Γαλλία και παρακαλώ πρώτα την κυρία Μαράτου Αλιπραντή να λάβει το λόγο για να μας κάνει την παρουσίασή της. Ευχαριστώ πολύ. Thank you ε, for me in this ε, Ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε στην ακρόαση αυτή. Στον με ιδιαίτερη τιμή και υπερηφάνεια για την ε, απόφαση σας αυτή, για την συζήτηση του θέματος αυτού, του, του διαφιλονικούμενου θέματος της, του τοκετού σε ανωνυμία. Η ιδέα του ποιος, ποιος είναι ο ρόλος του γονέα της, ε, σχέσεις της μητέρας με το παιδί του του παιδιού προσαρμόζονται σε διάφορους διαφορετικούς ε, κανόνες, πρακτικές, έθιμα που όμως έχουν ε, διαφιλονικούμενο περιεχόμενο. Τα προστρονομιοθωτικά συστήματα όμως στηρίζονται πάνω απ' όλα στην αυτόματη αναγνώριση της σχέσης της μητέρας με το παιδί από τον τοκετό και μόνο. Στην ε, Ελλάδα δεν υπάρχει δυνατότητα για ανώνυμο τοκετό, για τοκετό σε ανωνυμία. Με βάση τον αστικό κώδικα είναι υποχρεωτική αναγνώριση, η δήλωση μάλλον του, το, της γέννησης του παιδιού. Υποχρεώς ε, σε δήλωση του γέννησης είναι ο πατέρας εφόσον υπάρχει, ο, τρός με ευτήρας ή ΜΕΑ ή οποιοδήποτε άλλο των παρών κατά, την, κατά τον τοκετό. Αυτή η δήλωση πρέπει να λάβει χώρα μέσα στις 10 ημέρες από τον τοκετό και με ιδιαιτερότητα της ελληνικής νομοθεσίας η γυναίκα, η μητέρα δηλαδή είναι υποχρεωμένη η ίδια να κάνει τέτοια δήλωση αλλά μπορεί να αποστείλει εκπρόσωπο με συμβολιογραφικό πληρεξούσιο. Έτσι λοιπόν, αντίθετα με άλλε ευρωπαϊκέ χώρε όπω η Γαλλία, η Αυστρία, το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο, δεν γνωρίζει στο νομοθετικό τη σύστημα τον τοκετό σε ανωνυμία. Έτσι λοιπόν και η εγκατάλειψη νεογνού στο νοσοκομείο θεωρείται και παράβαση του νόμου και ποινικό αδίκημα. Δεν μπορεί κανεί δηλαδή να εγκαταλείψει το παιδί του στο νοσοκομείο όπω σε άλλε χώρε. Τη Σλοβακία, όπω είπατε. Στην περίπτωση επίση του της υιοθεσίας εφαρμόζεται η αρχή του απορρίτου των στοιχείων και με βάση την πρόσφατη νομοθεσία η γονική συνένεση μπορεί να χορηγηθεί κατόπιν ε, δικαστικής αδείας, αυτή είναι η πρόσφατη νομοθεσία του 2008, πάντοτε το παιδί μπορεί να αναζητήσει τους ε, φυσικούς του γονείς μετά την ενηλικίωση από τα 18 του και μετά. Τώρα, και αντίθετα με αυτά που σας είπα, στη Γαλλία, την Αυστρία, το Λουξεμβούργο εφαρμόζεται διάκριση μεταξύ του, της βιολογικής και της νομικής μητρότητας. Δηλαδή μια μη ύπανδρη μητέρα δεν θεωρείται αυτόματα μητέρα του παιδιού της επιτρέπει ο νόμος δηλαδή να παραμείνει επισήμως άγνωστον στοιχείων και τι είναι η φυσική μητέρα του παιδιού η νομοθεσία στη Γαλλία αναφέρεται στον τοκετό υπό χ όνομα άγνωστο δηλαδή και επιτρέπει σε μια μητέρα να, ε, να προχωρήσει το τοκετό χωρίς να αποκαλύψει ταυτότητά της προσφέρεται δε η ατροφαρμακευτική περίθελψη και η μέρημνα που απαιτείται όπως άλλωστε συμβαίνει και στην Αυστρία η μητέρα έχει το δικαίωμα μέσα σε 8 εβδομάδες να ε, διεκδικήσει το παιδί της πριν αυτό διατεθεί σε υιοθεσία, αλλά παραμένει ασαφές, ασαφής η προέλευση του νόμου αυτού κατά πάσα πιθανότητα στόχο είχε να προστατεύσει τις γυναίκες σε περίοδο πολέμου και να τους επιτρέψει να ε, φέρνει το παιδί τους στη ζωή ανώνυμα, όμως όχι κατά πάσα πιθανότητα και να διευκολύνει τις υιοθεσίε. Τώρα έχουμε περίπου 600 γυναίκες στην ε, Γαλλία, εκ των οποίων 10% ανήλικες, το χρόνο που κάνουν χρήση του δικαιώματος αυτού. Περιορισμένος λοιπόν ο αριθμός αυτές τις 600 γυναίκες ε, αν συγκριθεί δε με τις 10.000 το χρόνο που είχαμε στη δεκαετία του 80. Πρόσφατη μεταρρύθμιση της γαλλικής νομοθεσίας επίσης δίνει τη δυνατότητα στη μητέρα να προσφέρει στοιχεία για την ταυτότητά της Προσωπικέ πληροφορίες σε σφραγισμένο φάκελο τον οποίο θα ζητήσει, ο θα ζητήσει να χορηγηθεί στο παιδί τη όταν αυτό είναι ηλικιωθεί χωρίς όμως να είναι υποχρεωτικό να δώσει τέτοια στοιχεία να δώσει δηλαδή την, ε, την ιστορία της την προσωπική. Λέγεται επίσης ότι το σύστημα αυτό σαν στόχο έχει να προστατεύσει τη μητέρα όταν αυτή προστιμά την ε, μόνιμη, την επαόριστον ανωνυμία και όχι την ε, γνωστοποίηση των στοιχείων της. Στη Γερμανία και την Ελβετία τώρα. Στη Γερμανία υπάρχουν τρεις προτάσεις για τη θέσμιση, θέσπιση το κετού σε ανωνυμία γιατί υπάρχει μια ιδιαίτερη έμφαση στον αδιάρρηκτο δεσμό γονέων και παιδιού ε, στο γερμανικό οικογενειακό δίκαιο. Και επίσης στη Γερμανία όπως και στην Ελβετία εξασφαλίζεται από το Σύνταγμα αυτό το αυτή η δυνατότητα. Στην Ιταλία δεν προβλέπεται υποχρέωση για τη μητέρα να ε, δώσει τα στοιχεία της, όπως άλλωστε συμβαίνει και στο Βέλγιο, όπου όμως υπάρχει δυνατότητα για τον τοκετό σε, στοιχεία, σε συνθήκες ανωνυμίας, με τη δυνατότητα όμως και για το παιδί αργότερα να αναστήσει τα στοιχεία του και τη γενιά του. Οι γυναίκες έχουν διεκδικήσει το δικαίωμα για το κετό σε ανωνυμία και έχουν προκαλέσει πολλές συζητήσεις τα τελευταία δέκα χρόνια στην Ευρώπη και στη Γαλλία ιδιαίτερως. Υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι υποστηρίζουν το σύστημα και θέλουν να ενισχυθεί η νομοθεσία. Υπάρχουν όμως και εκείνοι που αντιτίθενται στο σύστημα αυτό και στην πρακτική αυτή. Για να καταλάβει κανείς ε, το πλαίσιο του δημόσιου διαλόγου θα ήθελα να παρουσιάσω τώρα τα επιχειρήματα των δύο πλευρών. Πρώτο επιχείρημα λοιπόν να αποτρέπονται η ε, εγκατάλειψη έκθεση παιδιού. Αυτή η ιδέα του έκθετου παιδιού έχει να αποτρέπεται η εγκατάλειψη, η έκθεση παιδιού, αυτή η ιδέα του έκθετου παιδιού έχει να κάνει με την ιστορική πορεία που έχουμε από τις αρχές του 20ου αιώνα. Ε, υποστηρίζουν λοιπόν ε, αυτοί που είναι υπέρ του το και του ανωνυμία ότι διευκολύνεται η δυνατότητα της υιοθεσίας και μειώνονται οι περιπτώσεις μια γυναίκα να εγκαταλείψει το παιδί της. Άρα, ένα τέτοιο μέτρο θέσουσε και τη μητέρα και το παιδί. Από την άλλη, εάν η εγκατάλειψη λάβει χώρα σε μεταγενέστερο στάδιο, το παιδί δεν μπορεί να υιοθετηθεί εγκαίρως Μειώνεται δηλαδή και ο αριθμός των διαθέσιμων για υιοθεσία παιδιών. Μια θετική λοιπόν ε, πτυχή θα ήταν η επιτάχυνση των διαδικασιών της υιοθεσία που θα ήταν βέβαια προς το συμφέρον των παιδιών ιδιαίτερος, αν και αμφισβητείται ένα τέτοιο αποτέλεσμα, γιατί δεν είναι βέβαιο ότι ένα τέτοιο σύστημα δεν ε, αμφισβητείται το κατά πόσο ένα τέτοιο σύστημα το κετού ανωνυμία θα εξαφάνισε τελείω τι πιθανότητε φώνευση του παιδιού, του νεογνού δηλαδή αμέσω μετά το κετό ή της εγκατάλειψης του. Επίσης μια άλλη επιχειρηματολογία είναι ότι η τη εγκαταλειψη του επιση μια να ελέγχει η ίδια το κορμί της και την, τον ιδιωτικό βίο. Πρέπει λοιπόν το σύστημα, όπως ζητούν ορισμένοι, να διατηρηθεί αλλά με ορισμένους περιορισμούς και να είναι συμπληρωματικό το και σε ανωνυμία ως προς την λυπή νομοθεσία. Και άρα μπορεί να αποτελέσει επέκταση του δικαιώματος της εθελούς, του εθελούσιου τερματισμού εγκυμοσύνης, της άμπλουσης δηλαδή μια γυναίκα μπορεί να είναι σε θέση να αρνηθεί τη μητρότητα, ιδιαίτερα αν έχει πέσει θύμα ε, βιασμού ή ε, άλλης μορφής βίας σχετικής. Ε, αυτό βέβαια είναι το επιχείρημα των φεμινιστριών. Αγνοεί όμως το βιολογικό δεσμό και τον κοινωνικό δεσμό. Πρόκειται για μια θέση την οποία έχουν υιοθετήσει και οι γονείς φετών παιδιών, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι είναι πιο ισχυρή κοινωνική παρά βιολογική δεσμοί. Η ομιλήτρια ομιλεί πάρα πολύ γρήγορα και είναι αδύνατο να την παρακολουθήσουν οι διερμηνείς. Προσπαθούμε λοιπόν με τα επιχειρήματά μας να εξηγήσουμε και την βιολογική αλλά και την κοινωνική διασύνδεση του παιδιού με την οικογένειά του. Στη Γαλλία επικρατεί η αρχή του δικαίου του εδάφους, γιους σόλης, αντί για το γιους ε, σάνγκουις, αντί για το δίκαιο δηλαδή του αίματος ως προς την ε, κληρονομιά, ως προς την πορεία μάλλον ενός ανθρώπου μέσα στην οικογένειά του. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι αγωνίζονται για την κατάργηση του συστήματος αυτού στις Γαλλία, στην ε, τοκετό σε ανωνυμία, διότι παραδείγματι δεν επιτρέπεται στο παιδί η αναζήτηση της γενεάς του, ε, αισθάνεται την εγκατάλειψη, κόβονται οι ρίζες του παιδιού. Στην ε, Γαλλία, ύστερα από δεκαετία τέτοιων συζητήσεων και από πολυάριθμες αναζητήσεις της γενιάς ανθρώπων που είχαν εγκαταλειφθεί από τις μητέρες τους. Επανήλθε το θέμα αυτό. Και υπάρχει μία τάση για την ενίσχυση της υιοθεσία incognito, χωρίς δηλαδή διατήρηση των στοιχείων της γενιάς. Αυτό το έχει ακολουθήσει και η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχουν επίσης αλλαγές και στις κοινωνικές προδιαγραφές και την κοινωνική συμπεριφορά στην Ευρώπη, όπως γνωρίζουμε από, χάρη στα στατιστικά και τα δημογραφικά μας στοιχεία. Είναι πολύ χαμηλότερη ε, τα ποσοστά των ε, θανατώσεων νεογνών, μικρότερα τα ποσοστά των ε, εφήβων μητέρων, ε, αύξηση των ποσοστών και αποδοχή βέβαια των εξωγαμιαίων τοκετών στην Ευρώπη. Συγκρινόμενη δε με το 8% το 1975 έχει αυξηθεί ιδιαίτερα αυτή η αναλογία. Επίσης η συμβίωση έχει αντικαταστήσει πολύ συχνά το γάμο. Πολλά από τα ζευγάρια είναι μόνο σε συγκατοίκηση όταν γίνεται το πρώτο τους παιδί και όχι παντρεμένα. και αποκόπτεται η σχέση της ε, μητρότητας, της πατρότητας από τον γάμο, το θεσμό του γάμου. Έχει αλλάξει λοιπόν η κοινωνική συμπεριφορά στην Ευρώπη. Για να προχωρήσουμε προς τα συμπεράσματα, υπάρχουν πολλοί λόγοι που οδηγούν, οδήγησαν μάλλον στη θεσμοθέτηση της, ε, του απόρριτου του κετού, στη δεκαετία του 50, που τώρα όμως πλέον δεν έχουν λόγο ύπαρξης. Χώρες που γνωρίζουν το σύστημα αυτό και θα ήθελαν να το καταρκήσουν θα μπορούσαν να εισαγάγουν μια υποχρεωτική διαδικασία χάρη στην οποία θα ήταν σε θέση το παιδί ενηλικιούμενο να διεκδικήσει την ενημέρωση για τα στοιχεία των γονιών του. Υποχρεωτικό λοιπόν αυτό. Βέβαια υπάρχουν άλλα επιχειρήματα που δύσκολα μπορεί κανείς να συμφιλιώσει με Ταξί να συγκεράσει δηλαδή δικαιώματα της μητέρας, το προσωπικό της βίος, το απόρριτο, δικαιώματα του παιδιού στο να γνωρίσει τη γενιά του, δικαιώματα των θετών γονιών. Πλην όμως όταν υπάρχει η δυνατότητα, μάλλον όταν υπάρχει η νομοθετική επιταγή το παιδί να είναι σε θέση να ανέβρει τους φυσικούς του γονείς, νομίζω ότι αυτή θα πρέπει να επικρατεί τον λοιπόν. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Επίσης, Υπάρχει ε, μία σειρά θέσεων η οποία προτείνει την πολυγονεϊκότητα, pluriparentalite δηλαδή να υπάρχει δυνατότητα να αναγνωριστεί πολλαπλός δεσμός του παιδιού με περισσότερα του ενός πρόσωπα, μητέρας ή πατέρες. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μια, μια λύση. Αυτή ήταν η παρέμβασή μου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για αυτή την παρουσίαση. Και τώρα να δώσω το λόγο στη Μαρή Ζωζέ Κελέρ, η οποία πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τέρων στο Παρίσι. Μεών στο Παρίσι. Ευχαριστώ κύριε και κύριοι. Ευχαριστώ καταρχάς να συστηθώ. Είμαι η Μαρή Ζωζέ Κελέρ, πρόεδρος του Εθνικού Συλλόγου Μεών της Γαλλίας στο Παρίσι και σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε για αυτή την ακρόαση. Είναι τιμή για μένα και για, την, για τον κλάδο των μεών να έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε εδώ για την πείρα μας σε σχέση με το θέμα των τοκετών σε ανωνυμία. Είναι ένα θέμα που για μένα είναι ιδιαίτερα σημαντικό και προσφυλές, διότι ως ΜΕΑ έχω ιδιαίτερη εμπειρία από τέτοιους τοκετούς και γυναίκε που έχουν γεννήσει σε ανωνυμία. Mm. Ποιοι είμαστε πρώτα απ' όλα. Ο Σύλλογο των ΜΕΟΝ είναι η αρμόδια αρχή για την καταγραφή, τη ρύθμιση και τον έλεγχο καθώς και την επαγγελματική άσκηση του επαγγελματο. της ΜΕΑ στη Γαλλία και επίσης ε, προστατεύεται την ε, δεντολογία του επαγγελματο Μιλάμε για ένα σύλλογο όπου ανήκουν υποχρεωτικά όλες ε, οι ΜΕΕ με επαγγελματική άδεια να ξεσκούν το επάγγελμα αυτό, 20.000 περίπου στη Γαλλία. στοχο είναι η υπεράσπιση και η διασφάλιση της δημόσιας υγείας ό,τι αφορά τις γυναίκες και τα νεογνά. Να σας πω με λίγα λόγια πώς έχει κατάσταση στη Γαλλία σε ό,τι αφορά τον τοκετό σε ανωνυμία. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τους τοκετούς σε ανωνυμία, η Γαλλία αποτελεί εξαίρεση στην Ευρώπη κατά τρόπο διτό. Πρώτα απ' όλα γιατί λόγω της ιστορίας της πρακτικής αυτής η Γαλλία έχει μακρά παράδοση τοκετών σε ανωνυμία. Από τον 17ο αιώνα είχε προβλεφθεί σύστημα εγκατάλειψης ε, των ε, βρεφών και έπειτα προβλέφθηκε από το νόμο από τη Γαλλική Επανάσταση το 1793 ο τοκετός σε ανωνυμία. Η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που έγινε έκτοτε ήταν το 2002. Άλλη ιδιαιτερότητα της Γαλλίας είναι ότι είναι μια χώρα που διασφαλίζει στις γυναίκες το υψηλότερο βαθμό προστασίας, ε, απορρίτου και ταυτότητα επίση, Προστασία τη ταυτότητά τους. Θα το δούμε και κατόπιν. Τώρα, τι είναι ο τοκετός σε ανωνυμία. Είναι ο τοκετός που επιτρέπει σε μια γυναίκα να παρακολουθείται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της και να γεννήσει δωρεάν, είτε είναι ενήλικη είτε όχι, είτε είναι ύπανδρο ή όχι, είτε είναι γαλλική υπηκότητα ή αλλοδαπή δεν είναι υποχρεωμένη να αποκαλύψει την ταυτότητά τη και μπορεί να λάβει τη διασφάλιση ότι η ταυτότητα αυτή δεν θα αποκαλυφθεί σε τρίτους χωρίς την δική της εξουσιοδότηση. Στόχοι. Στόχοι είναι να προστατεύσουμε την υγεία της μητέρας και του παιδιού, να αποφύγουμε του ε, τους τοκετούς, ε, τις, ε, τις διακοπές εγκυμοσύνης παρανόμως, επίσης την θανάτωση των νεογνών, και να παρακολουθήσουμε σωστά από υγειονομική άποψη την εγκυμοσύνη καθώς και τον τοκετό σε καλές συνθήκες υγεία και για τη μητέρα και για το παιδί και να προστατεύσουμε και τη σωματική ακαιρεότητα των μητέρων που μπορεί να απειλείται. Ποιε είναι οι συνέπειε τώρα. Για το παιδί θα υπάρχει επιστοποιητικό γέννηση κενό. Ε, το παιδί το αναλαμβάνουν αμέσως οι υπηρεσίες της κοινωνικής ε, προστασίας και ασφάλειας ε, για τα παιδιά με στόχο την υιοθεσία. Ενώ η μητέρα έχει μια προθεσμία δύο μηνών προκειμένου να αλλάξει άποψη γνώμη αν το θέλει και στη συνέχεια το παιδί γίνεται κινδεμονεύεται από το κράτος και η μητέρα δεν θα μπορεί πλέον να το ξαναδεί. Για τη μεταρρύθμιση του 2002 που ήταν ιδιαίτερα σημαντική. Τι την προέβλεψε η Σεγκολέν Ρουαγιάλ, η οποία ήταν υπεύθυνο υπουργό οικογένεια το 2001 και οδήγησε στο νόμο τη 22 Ιανουαρίου του 2002 που κύρωσε το σύνολο του Γαλλικού Κοινοβουλίου, τη Γαλλική Βουλή. Είχαμε εδώ ένα πλαίσιο διτό ε, της αυξανόμενες απαιτήσει των συλλόγων για τα παιδιά που είχαν ε, γεννηθεί ανώνυμα και των ε, μητερών αυτών που δεν είχαν αποκαλυφθεί τα στοιχεία τους, καθώς και τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού που είχαν ε, ετοιμαστεί από την ΟΗΕ ούτως ή άλλως από το 1999. Εκεί έπρεπε να αναγνωριστούν τα ειδικά δικαιώματα των παιδιών. Η, συνθήκη αυτή, η σύμβαση κυρώθηκε ούτως ή άλλως ε, από τη Γαλλία λίγο νωρίτερα και ορίζει η σύμβαση αυτή ότι στο μέτρο του δυνατού το παιδί έχει δικαίωμα να γνωρίζει τους γονείς του, την καταγωγή του. Κατόπιν, μετά από την ε, μεταρρύθμιση αυτή, οι τοκετής ανωνυμία επιτρέπονται και πάλι, αλλά τη στιγμή του τοκετού η μητέρα μπορεί να αποφασίσει εάν θα δώσει τα στοιχεία της, ε, του ιστορικού της για να μπορεί το παιδί να λάβει γνώση, ιδίω για την υγεία του, την υγεία του πατέρα του, τις συνθήκες γέννησής του, την καταγωγή του παιδιού και επίσης ενθαρρύνεται η μητέρα να αφήσει μια επιστολή ή ένα αντικείμενο το οποίο θα παραδοθεί στη συνέχεια στο παιδί. Επίσης η μητέρα καλείται σε σφραγισμένο φάκελο να αφήσει τα στοιχεία της ταυτότητάς της, όνομα τεπώνυμο και ημερομηνία γέννησης, στοιχεία τα οποία θα, θα περιλαμβάνονται ε, σε ένα φάκελο μαζί με το προτινόμενο ονοματεπώνυμο για το παιδί, όπως το δίνει η μητέρα, καθώς και το φύλλο, η ώρα, ε, η ημερομηνία και ο τόπος γέννησης. Ε, το φάκελο αυτό θα παραμείνει κλειστός εκτός εάν η μητέρα κάποια στιγμή αποφασίσει να άρει το απόλυτο, κατά τη διάρκεια της ζωής της. Αυτό οδήγησε στη δημιουργία του Εθνικού Συμβουλίου στην για την πρόσβαση στην προσωπική καταγωγή του ατόμου, την ΚΝΑΟΠ, η οποία επιτρέπει στα παιδιά που το επιθυμούν να αναζητήσουν τους γονείς τους. Και ε, χρησιμεύει ως διαμεσολαβητής μεταξύ γονέων και παιδιών. Ε, έχει αναλάβει το Συμβούλιο αυτό να συγκεντρώνει τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με τους τοκετούς σε ανωνυμία στην Γαλλία. Εάν το παιδί λοιπόν αναζητήσει στοιχεία για την καταγωγή του θα πρέπει υποχρεωτικά να απευθυνθεί στο Εθνικό Συμβούλιο πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία καταγωγή. Και αυτό ακριβώ το Συμβούλιο είναι που θα ξεκινήσει και θα εκκινήσει τη διαδικασία ανοίγματο του φακέλου ε, του παιδιού. Ποια στοιχεία τώρα είναι αυτά στα οποία μπορεί να έχει πρόσβαση ένα παιδί. Ο εκπρόσωπο του Εθνικού Συμβουλίου μπορεί να αποκαλύψει τις εξής πληροφορίες, αυτές που δεν είναι σε σφραγισμένο φάκελο, πληροφορίες που κάποιες φορές αρκούν στο παιδί για να μπορέσει να χτίσει την ταυτότητά του. Όσον αφορά τα στοιχεία της ταυτότητας της μητέρας υπάρχουν διάφορες δυνατότητες. Πρώτον, η μητέρα μπορεί να έχει αρνηθεί να αποκαλυφθεί η ταυτότητά της, κάτι που συμβαίνει περίπου στο 40% των περιπτώσεων, οπότε σε αυτή την περίπτωση το παιδί έχει δεν έχει καμία πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου. Εάν η μητέρα όμω έχει αφήσει τα στοιχεία τη στο φάκελο, το Εθνικό Συμβούλιο θα έρθει σε επαφή μαζί τη ε, μυστικά και θα ρωτήσει εάν συμφωνεί, εάν συγκατατίθεται προκειμένου να έρθει το απορρίτω. Σε αυτήν ε, τη χρονική στιγμή η μητέρα μπορεί να αποδεχτεί να αρνηθεί βεβαίω και γνωρίζουμε ότι περίπου 40% των μητερών αποδέχονται, αποδέχονται να έρθει το απορρίτω είναι λοιπόν μειονότητα σε κάθε περίπτωση. Ο ρόλος των νέων είναι καθοριστικός στην παρακολούθηση των γυναικών που ε, ε, γεννούν παιδιά σε ανωνυμία πρώτα απ' όλα συνδράμουν τις γυναίκες, ε, συνεργάζονται με τις κοινωνικές υπηρεσίες για την προστασία των παιδιών και το Εθνικό Συμβούλιο για την πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία καταγωγής, αναλαμβάνει τη σύνταξη του φακέλου για το κάθε παιδί και συμπληρώνει και τον ιατρικό φάκελο καθώς και το βιβλιάριο υγείας των παιδιών, εξασφαλίζοντας βεβαίως την ανωνυμία της μητέρας. Η ψυχολογική παρακολούθηση είναι επίσης εδώ πολύ σημαντική, διότι πρέπει να γίνεται με πλήρη σεβασμό των επιθυμιών και των αναγκών της μητέρας. Δεν μπορεί να μιλά κανείς ποτέ για εγκατάληψη, αλλά για υιοθεσία. Η μητέρα θα πρέπει να μπορεί να επιλέξει το όνομα τεπώνυμο και αν αρνηθεί να το κάνει θα πρέπει η νέα να προτείνει ένα όνομα τεπώνυμο. Επίσης η μητέρα θα πρέπει να μπορεί να κρατήσει για λίγα λεπτά στην αγκαλιά της το παιδί, να έχει λίγα λεπτά ε, μόνοι μαζί του και στη συνέχεια θα πρέπει να τύχει περίθαλψη σε, ένα ειδικό, σε μια ειδική υπηρεσία στο νοσοκομείο, όχι αυτήν ε, των τοκετών ε, και να μπορεί να είναι σε επαφή και με άλλες γυναίκες που μόλις έχουν γεννήσει. Πρέπει να πούμε ότι τη δεκαετία του 70 είχαμε τουλάχιστον 10.000 γεννήσεις σε ανωνυμία πριν την απελευθέρωση των κεφαλών διακοπών κοίησης. Τώρα έχουμε, περισ... έχουμε ακόμη περισσότερες γεννήσεις στη Γαλλία. Ποιες είναι οι πιο συνηθισμένες περιπτώσεις. Είναι οι πολύ νεαρές μητέρες οι οποίες ζουν μόνες εκτός οικογενειακού πλαισίου και συνήθως είναι κάτω των 25. Επίσης πολύ συχνά ανήλικες. Δεύτερη περίπτωση είναι οι γυναίκες οι οποίες προέρχονται από οικογένειες μουσουλμανικές. Ισλαμι... Ισλαμικές οι οποίες ζουν ακόμη στο σπίτι των γονιών τους και εκτός γάμου έχουν ε, μείνει έγκες οπότε μπορεί να τιμάσουν όπως θεωρούν οι οικογένειές τους την οικογένεια και να έχουν βεβαίως ε, να υποστούν δραματικές συνέπειες. Ναι. Μπορεί σε κάθε περίπτωση μπορεί να τις ξαναστείλουν στη χώρα τους μπορεί να τις οδηγήσουν σε εξαναγκαστικούς γάμους ή να δεχτούν και επίθεση προσωπική. Σύμφωνα με τον καθηγητή αριών της Ιατρικής Ακαδημίας της Γαλλίας, οι γυναίκες αυτές είναι περίπου το 50% των γυναικών στις μεγάλες πόλεις και 30% σε άλλες γεωγραφικές περιοχές στην επαρχία. Επίσης έχουμε γυναίκες που αντιμετωπίζουν σοβαρές ηλικίες δυσκολίες, είτε αρκετά νέες είτε και μεγαλύτερες ηλικίες. Υπάρχει ένα σημαντικό μερίδιο γυναικών που προέρχονται από οικογένειες με... μάλλον που προέρχονται από ε, που έχουν άνετη κοινωνική ζωή, αλλά παρόλα αυτά έχουν οικογενειακές πιέσεις προκειμένου να συνεχίσουν την επαγγελματική τους ούτω καθεξής. Επίσης οι γυναίκες θύματα βιασμών ή επίσης εκείνες που αρνούνται την εγκυμοσύνη τους. Ο λόγος τώρα που οδηγεί τις γυναίκες να γεννούν σε ανωνυμία μπορεί να είναι, οι λόγοι αυτοί μπορεί να είναι πολλοί. Πρώτα απ' όλα ηλικέ δυσκολίες για να συντηρήσουν το παιδί. Ε, οι γυναίκε αυτέ θεωρούν ότι αν δώσουν το παιδί για θεσία, του επιτρέπουν να έχει μια καλύτερη τύχη. Άλλε δεν είναι σε ψυχολογική κατάσταση να αναλάβουν ένα παιδί, διότι μπορεί να έχουν βιαστεί ή να έχουν ε, μείνει από ατύχημα. Επίση, οι γυναίκες αυτές που γεννούν σε ανωνυμία πολύ συχνά μπορεί να έχουν ε, ψυχολογικές δυσκολίες ή να βρίσκονται σε συνθήκες συναισθηματικής και κοινωνικής απομόνωσης. Μια πολύ μικρή αναδρομή στο τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αν και δεν είμαι ειδήμων και παρόλο που το θέμα το έχουμε εν μέρη θίξει, υπάρχουν ε, χώρες που επιτρέπουν την, τους τοκετούς ανωνυμία, αλλά όλες οι χώρες, πολλές χώρες μάλλον έχουν ε, κανόνες παρόμοιους με τις Γαλλίας. Η ένδειξη του ονοματεπονίμου της μητέρας του πατέρα είναι υποχρεωτική σε κάποιες ε, χώρες, ε, σε κάποιες χώρες της Ευρώπης, οπότε στη Γαλλία υποδεχόμαστε πολλές αλλοδαπές μητέρες, από το Βέλγιο, την Αλγερία επίσης, 15% του συνολικού αριθμού γυναικών που γίνονται σε ανεμία. Στη Λίλ, για παράδειγμα, ένα μεγάλο ποσοστό, το 30% περίπου των γυναικών που γίνονται σε ανεμία, προέρχονται από το Βέλγιο. Οι χώρε που επιτρέπουν ε, στι μητέρε να μην δίνουν τα στοιχεία του είναι η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, η Αυστρία από το 2001 και η Ουγγαρία. Οι χώρες που δεν επιτρέπουν το τοκετό σε είναι η Γερμανία, το Βέλγιο, η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η, η Ελβετία και παρόλα αυτά, ε, και υπάρχουν κάποιοι ενδιασμοί, η Ελλάδα, δεν θα τις αναφέρω έτσι κι αλλιώς όλες, αλλά υπάρχουν όπως έλεγα ενδιασμοί ε, σε σχέση με κάποιες χώρες ειδικά. Προβλέπουν δηλαδή οι χώρες αυτές μεταρρυθμίσεις προκειμένου να επιτραπεί ο ε, το και ανωνυμία. Μεταξύ άλλων, όπως είπατε και εσείς ε, κυρία Πρόεδρε, στη Σλοβακία, στη Γερμανία και στο Βέλγιο. Ε, νομίζω Μιλή, μιλήσαμε επίσης για τις θηρίδες, τις νεουνών που υπάρχουν σε χώρες οι οποίες δεν επιτρέπουν το στο σε ανωνυμία. Εδώ μιλάμε για τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ελβετία, το Βέλγιο και τη Σλοβακία. Όπως ε, σας είπαμε προηγουμένως, η αρχή μιας στηρίδας νεογνών είναι το μωρό πρέπει να μπαίνει σε μια θερμοκοιτή, να μπαίνει σε μια η οποία μπορεί να βρίσκεται σε μια, να έχει ένα διαφανές άνοιγμα ε, από τη μία πλευρά και να, δίνει, να, έχει, να υπάρχει πρόσβαση από τον ε, δρόμο ώστε να μπορεί σε πλήρη ανωνυμία να αφήσει το μωρό εκεί. Πάντω αυτό δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ιατρική περίθαλψη του στον νεογνώ ούτε στη μητέρα είτε πριν είτε μετά τον τοκετό. Οπότε δεν είναι ικανοποιητική λύση και οι συνέπειε για το παιδί είναι φυσικά χειρότερε από ότι για ένα νεογνώ που γεννήθηκε σε ανωνυμία. Δηλαδή το μωρό, εάν επιβιώσει, ουδέποτε θα μπορέσει να έχει πρόσβαση στα στοιχεία της καταγωγής του. Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν θα έλεγα ότι σε ό,τι αφορά τους τοκετούς σε ανωνυμία βεβαίως η Γαλλία αποτελεί εξαίρεση στην Ευρώπη γιατί ο τοκετός σε ανωνυμία ούτως ή άλλως είναι ένα ζήτημα αμφιλεγόμενο ε, και υπάρχουν εδώ δικαιώματα συμβίβαστα όπως το, ο σεβασμός της ελευθερίας επιλογής της μητέρας αλλά και το δικαίωμα του παιδιού να γνωρίζει την καταγωγή του. Αυτά αντιτίθεται μεταξύ τους. Ο ρόλος των νεών ήταν να προσπαθήσουν να παρέμβουν σε αυτή τη συζήτηση και τον συμβιβασμό μεταξύ των δικαιωμάτων των μητερών και των παιδιών. Πάντως, αυτή τη στιγμή, για τις γυναίκες είναι σίγουρο ότι δεν μπορούν να δημιουργήσουν συστηματικούς παιδιούς με, το, με τα παιδιά τους και αυτό που πρέπει να μας απασχολήσει είναι ότι δεν θα πρέπει να υπερισχύσουν τα δικαιώματα των μεν εις βάρος των δε και αντιστρόφως. Από την προσωπική μου εμπειρία είναι ότι το δικαίωμα αυτό επιτρέπει πραγματικά να ε, προστατεύσουμε τη ζωή και των μητέρων και των παιδιών και πραγματικά οι γυναίκε αυτές που αναγκάζονται να περάσουν σε τοκετό σε ανωνυμία είναι πραγματικά δυστυχισμένε. Δεν υπάρχει καμία που να μην κλαίει τη στιγμή του τοκετού. Αλλά θέλουν και η χειρονομία τους να έχει ένα νόημα. Θέλουν δηλαδή να δώσουν μια ευκαιρία στο παιδί. Ε, μια ευκαιρία να μπορέσει το παιδί να βρει μια οικογενειακή ιστία που να το αγαπά. Ε, να βρει ένα πατέρα και μια μητέρα. Να ε, βρει τελικά και να έχει τις υλικές συνθήκες που θα επιτρέψουν να μορφωθεί, να είναι σε καλύτερη κατάσταση από ότι η ίδια η μητέρα θα μπορούσε να το προσφέρει. Μπορεί λοιπόν να σας φαίνεται παράξενο, αλλά ο τοκετός ξανωνυμία, καθώς και η θέση υιοθεσία ενός ε, νεογνού μπορεί να είναι και μια πράξη αγάπης από την πλευρά μιας μητέρας. Εάν θέλετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας για περισσότερες ε, πληροφορίες, ο ιστότοπος του Εθνικού Συλλόγου των Μεών της Γαλλίας είναι αυτός που βλέπετε στις οθόνες σας. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Um, uh, Ευχαριστούμε πολύ, λέει η Πρόεδρος. Και τώρα θα ακολουθήσει συζήτηση. Επιτρέψτε μου πρώτα πρώτα να δώσω στην κυρία Μπράιερ το λόγο, η οποία είχε την ε, πρωτοβουλία για αυτή τη δημοσιοκράση. Έχετε το λόγο κύριε Μπράιερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ιδιαίτερα σε ευχαριστώ τις δύο ομιλήτριες ήταν πολύ ενδιαφέρουσες, ενημερωτικές πλήρεις οι παρουσιάσεις τους. Η ιδέα για την ακρόαση αυτή προέκυψε από μια κατάσταση που αντιμετωπίζουμε στη Γερμανία, όπως είπατε και εσείς. Δεν είναι νομιμοποιημένη η ε, δυνατότητα του τοκετού σε στη Γερμανία. Κάνατε εσείς ε, λόγο ήδη για το δικαίωμα της αναζήτησης της γενιάς για το παιδί, το κάνατε λόγο για τα δικαιώματα των γυναικών, των μητέρων δηλαδή, αλλά υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα, ότι αν το παιδί δεν επιβιώσει, δεν υπάρχει το δικαίωμα της αναζήτησης της ε, γενιάς. Εδώ υπόλοιπον έχουμε να κάνουμε μια αντίφαση. Αυτό που με εντυπωσιάζει εμένα με τη Γερμανία είναι ότι θεωρείται, παρότι δεν υπάρχουν στι συγκεκριμένε στατιστικέ, ότι υπάρχουν περίπου αντίστοιχα ποσοστά με αυτά τη Γαλλία, δηλαδή 600, 600 το και στη Γερμανία το χρόνο, αλλά πολλοί από αυτού οδηγούν σε θανάτωση του νεογνού, διότι η μητέρα δεν έχει άλλη λύση, διότι η ίδια η θηρίδα νεογνών δεν την τη προσφέρει ικανοποιητική λύση. Υπάρχει κάμερα Φερρυπίν και μπορεί να αναγνωριστεί ταυτότητά τη. Δεν είναι ασφαλή ότι θα αφήσει εκεί το παιδί τη χωρί να αντιμετωπίσει προβλήματα μετά. Και πάνω απ' όλα ότι η γυναίκα δεν έχει καμιά βοήθεια στον τοκετό. Έχει υποστεί μεγάλη ταλαιπωρία. Έχει γεννήσει μόνη της η γυναίκα με κίνδυνο και της υγείας της, με φρικτές υγειονομικές συνθήκες φαίνεται από τι λένε οι γιατροί ότι τα στοιχεία είναι αντίστοιχα με αυτούς τους τοκετούς στην ε, Γαλλία, τους 600. Μιλούν λοιπόν οι γιατροί για 600 περίπου τέτοιους τοκετούς. Από αυτού τα στοιχεία που έχουμε είναι 25 περίπου θάνατοι νεογνών, θανατώσεις καλύτερα νεογνών και 25 νεογνά που υποτίθενται στην κοιτίδα. Για τα λοιπά όμως τα νούμερα, τα υπόλοιπα νούμερα μέχρι τον αριθμό των 600 είναι σκοτεινά. Δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί. Βέβαια υπάρχει ευρύτερο προβληματισμό για το ζήτημα αυτό μέσα στη Γερμανία μα έχει απασχολήσει το πρόβλημα και τη αναζήτηση τη γενιά για το παιδί, αλλά από την άλλη, αν θέλετε, πρέπει να το δούμε και ω δικαίωμα στη ζωή του παιδιού. Γιατί αν κινδυνεύει με θανάτωση σε περίπτωση που δεν υπάρχει αυτή η ανωνυμία σαν νομοθετική λύση, το παιδί τι, τι, τι δικαίωμα να έχει την αναζήτηση τη γενιά. Επίσης αυτό που με σοκάρει ιδιαίτερα είναι ότι υπάρχει μεγάλο ποσοστό γυναικών στη Γαλλία, κατά 50 μάλλον εκατό που γεννούν σε ανωνυμία, σε συνθήκε ανωνυμία, που προέρχονται από μουσουλμανικές οικογένειε, το οποίο δείχνει ότι τη σώζουμε τις ίδιες τις μητέρες από ίσως και σίγουρο θάνατο, από πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα εν πάση περιπτώσει στην οικογένειά τους. Μην ξεχνάμε ότι στη Γερμανία έχουμε τεράστιο πρόβλημα με τους ε, φόνους γυναικών για λόγους τιμής από μέλη της οικογένειάς τους. Ε, έτσι λοιπόν ερωτώ και εσείς προσωπικά τι είδους λύσεις μπορούσατε να προβλέψετε, δυνατότητα ενδεχομένω για μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία στο θέμα αυτό, γιατί και εμείς θα θέλαμε να εξασφαλιστεί μια δυνατότητα αντίστοιχη λύσης για όλες τις γυναίκες της Ευρώπης. Γιατί έχουμε να κάνουμε με το δικαίωμα της γυναίκας στη σωματική, στην, υγεία της, προσωπική της υγεία. Είναι δικαίωμα στην υγεία λοιπόν και νομίζω ότι αυτό θα μπορούσαμε να το υπαγάγουμε νομοθετικά σε μια νομική βάση που μιλάει για την υγεία. Γιατί αφαιρείται, αποστερείται από τη γυναίκα το δικαίωμα στην υγεία της, τη σωματική. Και επίσης, άλλωστε πρέπει να επισημάνω ότι είχα ζήσει, ήμουν παρούσα και σε μια ε, ακρόαση αντίστοιχη στη Γερμανία όπου ομίλησε η κυρία Κέσμαν, η προσκεκλημένη που δεν μπόρεσε σήμερα να έρθει δυστυχώς, η οποία μίλησε για το ζήτημα της κοινωνικής αποδοχής μιας γυναίκας ή μη αποδοχής καλύτερα μιας γυναίκας η οποία έχει γεννήσει σε συνθήκες ανωνυμίας. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να πω ότι κοινωνικά Στι δικέ μα κοινωνίε τώρα μπορεί να είναι αποδεκτό μια γυναίκα να έχει κάνει τρει, τέσσερι ή πέντε αμβλώσει ακόμη. Αλλά το να έχει γεννήσει τρία ή τέσσερα ή πέντε παιδιά και να τα έχει γεννήσει σε συνθήκε ανωνυμία και να τα έχει παραδώσει για υιοθεσία δεν είναι κοινωνικά αποδεκτό. Ερωτώ λοιπόν, γιατί αυτά τα διπλά μέτρα και σταθμά στην κοινωνία μας. Σε τι οφείλεται αυτό. Έχουμε μια κοινωνική αποδοχή αφενός της γυναίκας. Αφετέρου δε έχουμε ε, απόλυτη απόρριψη της γυναίκας που θέλει να γεννήσει σε συνθήκες ανωνυμίας ή που αφήνει το παιδί της σε μια κοιτίδα ή που το δίνει για υιοθεσία. Πού οφείλεται αυτό και πώς μπορούμε ενδεχομένως να το αντιμετωπίσουμε. Η Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μπράια. Κύριε Γκρένα. Ευχαριστώ πολύ. Δύο σύντομες ερωτήσεις μόνο, συμπληρωματικές. Και μία παρατήρηση ότι με γεμίζει αισιοδοξία το γεγονός ε, που αναφέρατε για τον περιορισμό, τη σημαντική μείωση των αριθμών γεννήσεων σε συνθήκες ε, ανωνυμίας, το κετών σε συνθήκες ανωνυμίας στη Γαλλία. Είναι ενθαρρυντικό αυτό και ένα πολύ σημαντικό μήνυμα ασφαλώς και για τα λοιπά ευρωπαϊκά κράτη. Για να τους δείξουμε ότι αν έχουν ανοιχτό πνεύμα και ε, νομοθεσία ανοιχτή, θα χρησιμοποιήσουν τη δυνατότητα αυτή μόνο οι γυναίκες που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Τουλάχιστον εγώ έτσι θα βλέπω τα πράγματα. Και επίσης γι' αυτό ερωτώ τι είδους πρωτοβουλία, όπως άλλωστε είπε και η συνάδελφος κυρία Μπράιερ, τι είδους πρωτοβουλία θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε στην κατεύθυνση αυτή και δεύτερη ίσως πιο άμεση ερώτηση υπάρχει κάποιος ευρωπαϊκός οργανισμός, ένωση, σύνδεσμος που ενδεχομένως οργανωτικά να μπορεί να προσφέρει υποστήριξη και στον οποίο ενδεχομένω και εμείς να μπορούμε να προσφέρουμε υποστήριξη ή εσάς να μπορούμε να σας υποστηρίξουμε και πολιτικά βεβαίως γιατί ιδιαίτερα με ενδιαφέρει η γυναίκα να μην αισθάνεται φόβο, να μην υφίσταται πιέσει στι συνθήκε αυτέ που αντιμετωπίσει και ίσω θα ήταν καλό και στην Γερμανία ιδιαίτερα να αναζητήσουμε την ενημέρωση για το τι συνθήκε επικρατούν, τι στοιχεία συλλέγονται, ποια είναι η κατάσταση σχέση με αυτές τις κοιτίδες ε, απόθεση νεογνών, διότι δεν είναι ικανοποιητική κατάσταση, πρέπει κάτι να αλλάξουμε. Έχει γίνει μόνο μισό βήμα θα έλεγα. Δεν έχει επιληθεί το πρόβλημα. Και θα ήθελα να εξασφαλιστεί δυνατότητα για τις γυναίκες να προσφέρεται ο τοκετός σε συνθήκες ανωνυμίας με ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και μέσα σε κλινικό περιβάλλον, σε συνθήκες υγειονομικές σωστές. Αυτό λοιπόν, αν έχετε κάποιες ιδέες να μας προσφέρετε, κάποιες υποδείξεις, πολύ ευχαριστώ να τις ακούσουμε. Ευχαριστώ πολύ, λέει η πρόεδρο κυρία η κυρία Στρέλα. Ευχαριστώ Πρόεδρα και εγώ ήθελα να ευχαριστήσω τις δύο προσκεκλημένες για τις πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες τους και τις παρουσιάσεις τους. Πραγματικά εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα θέμα αμφιλεγόμενο. Έχει να κάνει με θεμελιώδη δικαιώματα. Παρόλα αυτά μοιάζει προφανές ότι υπάρχουν πλέον ε, πλεονεκτήματα και για, τα, για τις μητέρες και για τα παιδιά. Ιδίως ό,τι έχει να κάνει με τις παράνομες ε, διακοπές κοίησης ή τις εγκαταλείψεις βρεφών και ούτω καθεξής. Παρόλα αυτά, στηρίζω λοιπόν την ιδέα ότι θα έπρεπε να υπάρχει νομοθέτηση και νομοθετική πρόνοια για το θέμα αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενδεχομένω. Και θα πρέπει να διακρίνουμε και μεταξύ διαφορετικών καταστάσεων. Λόγου χάρη. Διαφορετική είναι μια εγκυμοσύνη που προκύπτει από αιμομεξία, βιασμό ή άλλη άσκηση κατά μιας γυναίκας διότι εκεί είναι διαφορετικό το να θέλει κανείς να τρέξει σε το κετό σε ανωνυμία ή να απαγορεύεται, να μην επιτρέπεται η, η διακοπή κοίησης. Επίσης αναφέρθηκε και η περίπτωση των πολύ νέων μητέρων. Σε αυτή την περίπτωση δυσκολεύομαι να κατανοήσω γιατί πρέπει διαπαντός να χαθούν τα στοιχεία της ταυτότητας για το παιδί. Ενώ ότι σε αυτές τις περιπτώσεις με το πέρασμα του χρόνου μπορεί να αλλάξει η στάση της μητέρας. Μπορεί αυτό να προκύψει και με την ορίμανση του συγκεκριμένου ατόμου. Μόνο η ηλικία μπορεί να το προκαλέσει αυτό. Εάν θελήσει λοιπόν να αλλάξει γνώμη γιατί να αναμετάκλητο το μέτρο αυτό, γιατί να χάσει για πάντα το δεσμό με το παιδί. Νομίζω λοιπόν, εάν θέλουμε να προχωρήσουμε με μια νομοθετική πρωτοβουλία, να... θα πρέπει να σταθμίσουμε όλες αυτές τις διαφορετικές καταστάσεις. Ο Η περίπτωση των νεαρών μητέρων θα πρέπει σαφώς να διατηρήσει τη δυνατότητα της ανωνυμίας με τον σφραγισμένο φάκελο, με τα στοιχεία της ταυτότητας, τα οποία όμως θα πρέπει να παραμείνουν σφραγισμένα μέχρι λόγω χάρη την ενηλικίωση του παιδιού. Διότι και το παιδί, νομίζω, έχει δικαίωμα να γνωρίζει την ταυτότητά του. Και σήμερα, στη σημερινή εποχή, το δικαίωμα αυτό πρέπει να το προστατεύουμε όλο και περισσότερο, να διασφαλίζεται πάνω, πάνω απ' όλα. Δηλαδή να υπάρχει το δικαίωμα της ανωνυμίας των μητέρων εφόσον το επιθυμούν, αλλά να εγγυόμαστε και το δικαίωμα γνώσης της ταυτότητάς του από τον ίδιο το νέο, το μελλοντικό νέο δηλαδή το μωρό. Και οι νέες μητέρες, εάν αλλάξουν γνώμη, να έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν αυτό το δικαίωμα. Νομίζω λοιπόν η γαλλική περίπτωση όπου υπάρχει και ειδική επιτροπή συμβούλιο που ακούσαμε για την διατήρηση των στοιχείων της ταυτότητας που διασφαλίζει τόσο την καταγραφή όσο και την αποκάλυψη εφόσον χρειαστεί νομίζω είναι πολύ καλή αλλά και η μελλοντική ευρωπαϊκή νομοθεσία καλό θα ήταν να διακρίνει να διακρίνει μεταξύ των διαφορετικών αυτών περιπτώσεων που διαφέρουν πολύ μα πάρα πολύ μεταξύ τους. Ευχαριστώ. Ďakujem veľmi Ευχαριστούμε. Ε, θέλω να σα κάνω μια σύντομη παρατήρηση, κάτι το οποίο η κυρία Κέλλερ ανέφερε, για τι χώρε αυτέ που οποίες απαρίθμησε, όπου ε, θεσπίστηκε κάποιο νόμο όσον αφορά τι γεννήσει υπό καθεστώ και η Τσεχία όπως και η Σλοβακία έχουν τέτοιο νόμο όσον αφορά τις ε, τέτοιες ανώνυμες γεννήσεις ε, και αυτό να τρέξει το 2004 νόμος ο οποίος ισχύει. Όσον αφορά τώρα την ε, αρχιοθέτηση κάποιων πληροφοριών για τη μητέρα δεν ε, αναφέρεται το όνομα της μητέρας, ούτε το πιστευτικό ούτε και το μητρό αρένων ηθηλαίων. Το Επίσης υπάρχει κάποιος φάκελος με τα ιατρικά στοιχεία που σχηματίζεται εποφελία του ανηλίκου ούτως ώστε κατά τη διάρκεια της ζωής του όταν πάθει κάτι, όταν αρρωστήσει, εάν έχει κλινικό χαρακτήρα και χρειάζεται κάποιο είδου ε, μεταφορά, ο ασθενή να βοηθηθεί, <coughs> εφόσον υπάρχουν αυτά τα δεδομένα. Και δεν θα υπάρχει κάποιο ε, κίνδυνο για την υγεία του, η λήψη πληροφοριών. Πάντως ε, όλα αυτά τα στοιχεία Μόλις βγει από το νοσοκομείο η μητέρα, όλα αυτά τα δεδομένα υποβάλλονται στο Υπουργείο Υγείας. Φυλάσσονται εκεί και μόνο κατά την κρίση δικαστηρίου είναι δυνατόν να υπάρξει πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία. Μόνο, με δικαστική απόφαση επομένω αποκαλύπτονται αυτά τα στοιχεία. Εάν δεν θέλει να ζητήσει την προέλευσή του, ο ανήλικος όταν ενηλικιωθεί πια πάλι τότε απαιτείται από δικαστική απόφαση. Δεν αρκεί η επιθυμία του τόσο ώστε να βρει την άκρη. Θα πρέπει να υπάρχει συμφωνή με τη μητέρας και άρα γι' αυτό θα πρέπει οι αρχές να έχουν ε, κάποια στοιχεία για να μπορούν να βρουν τη μητέρα. Έχω πάντως ε, και εγώ κάποια εμπειρία στον αφορά τέτοιου είδους ε, ε, γεννήσεις, γιατί στη χώρα μου, την Σλοβακία, είμαι μέλος ενός τέτοιου υποπτικού οργάνου που βοηθά τις γυναίκες σε δύσκολες καταστάσεις και όσον αφορά την εγκυμοσύνη αλλά και όσον αφορά την τη, τη, τη βία κατοίκων, την οικογενειακή βία. Αυτός ο φορέας λειτουργεί εδώ και μία δεκαετία. Είχαμε 40 παιδιά που γεννήθηκαν από τις γυναίκες οργάνωσης. Ε, κάποια από αυτά τα παιδιά γεννήθηκαν υποκαθώς ανωνυμίας και ακολούθησε η υιοθεσία τους. Γι' αυτό σου λέω ότι από πρώτο χέρι ξέρω τι γίνεται με αυτό το θέμα. Έχουμε λίγο χρόνο, οπότε και τώρα θέλω να στραφώ στους εμπειρογνώμονες μας και αν μπορούν να απαντήσουν στα ερωτήματα. Έχετε το λόγο κύριε. Euh, πρώτα πρώτα να σας πω όσον αφορά την αναλογία των μουσουλμάν. Ε, δεν είναι το 50% στο Παρίσι και 30% στην υπόλοιπη Γαλλία σε σχέση με των γυναικών που γίνουν με αυτούς τις συνθήκες. Τώρα όσον αφορά την παρακολούθηση των γυναικών που έτσι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το συζητήσουμε γιατί μια γυναίκα που είναι έγκυος και η οποία βρίσκεται σε κάποια τέτοια ε, κατάσταση, βρίσκεται σε αδιέξοδο ε, όσον αφορά την εγκυμοσύνη, γεννά ε, σε συνθήκες μυστικότητας υπάρχουν κίνδυνοι πολλές φορές πρόκειται για πολύ νέες γυναίκες ακόμα δεν έχουν οριμάσει και μορφωθεί τα γεννητικά τους όργανα, πολλές φορές έχουν κάποιες ε, μοραγίες και επομένως υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι για σοβαρή βλάβη τη υγείας, οπότε αυτές ε, την χάνουν ιατρικής παρακολούθησης και μπορούν να κάνουν το τοκετό σε φυσιολογικές συνθήκες ο πλευράς ιατρικής όπως κάθε άλλη γυναίκα. Όντω, η Ένωση των Μεών μπορεί να συμμετάσχει σε κάποιε πρωτοβουλίες ώστε να προθεθεί αυτή η υπόθεση σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχει ήδη κάποιο τέτοιο φορέα που ονομάζεται European Midwife Association, EMA στα αγγλικά, Ένωση Ευρωπαίων Μεών και πρόκειται επομένω για ε, μια οργάνωση που εκπροσωπείται στην ε, Γαλλία και αν υπάρξει βοήθεια από τα ευρωπαϊκά όργανα μπορούμε να έρθουμε σε επαφή μαζί τους και μπορούμε έτσι να συνεργαστούμε προς την κατεύθυνση. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο να υπάρξει ε, σχετική νομοθεσία. Γιατί ακόμα και αν έχουμε 500 τέτοιες γεννήσεις ε, έχουμε 20 με 40 παιδιά τα οποία που ε, είναι παιδιά τα οποία άλλοτε και άλλοτε όχι. Γι' αυτό σου είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ κυρία Κέλλα. Μιλήσαμε για αυτές τις ε, τους στοκετούς υπό ανωνυμία, υπάρχει κάποια συγκράτηση των ποσοστών. Ε, υπάρχει όμως και κάποια μείωση των ε, εγκυμοσυνών. Κοιτάξτε, στη Γαλλία έχουμε 2,2 παιδιά ένα γυναίκα, επομένως θα πάμε καλά ε, δημογραφικού. Και έχουμε για διάφορους λόγους για τους οποίους έχουμε συρρήκνωση τέτοιου είδους γεννήσεων. Και αυτό γιατί, γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κάλυψη κοινωνική όσον αφορά αυτές τις ε, γυναίκες που βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Υπάρχουν κάποια τέτοια ιδρύματα, τις προστηρίζουν μέχρι να γίνει το παιδί ενός, ε, τις ε, βοηθάνε να βρουν δουλειά και έτσι να μπορέσουν να αρχίσουν κάποια επαγγελματική ε, καριέρα. Όμω αυτέ οι οποίε απειλούνται απειλούνται, να, να, να υποστούν κάποιο έγκλημα τιμή. Ε, αυτές τι περιπτώσεις πάντοτε υπάρχουν και αυτέ συνεχίζουν να θέλουν να γεννήσουν υποκατάσταση, υποκαθεστώς ανωνυμίας. Κύριε Παναγιώτοπουλη, το λόγο. Euh, remercier les euh, oratrices euh, de cette ήθελα να ευχαριστήσω τις ε, ομιλητρίες αυτή τη σημαντική ακρόαση και όσους, όσες μάλλον είχαν την πρωτοβουλία της. Είναι πολύ σημαντικά τα θέματα που καλύφθηκαν μας συγκλονίζουν οι ιστορίες που διαβάζουμε καμιά φορά για έκθετα στις ε, εφημερίδες ή για αφρικαλώτες πολλές φορές έχει διαπράξει η για που πολλες φορες εχει ότι υπάρχει η λοιπόν το γεγονός ότι υπάρχει περίθαλψη για τη μητέρα σε χώρες όπως η Γαλλία είναι πολύ σημαντικό. Είναι παράδειγμα που θα πρέπει να ακολουθήσουν και τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Και ιδιαίτερα με δεδομένο ότι προσφέρεται η δωρεάν ιατρική παρακολούθηση του, του, της εγκυμοσύνης και του τοκετού. Αυτό νομίζω είναι το βέλτιστο που θα μπορούσε να προσφέρει στον άνθρωπο η Γαλλία. Γιατί το να βοηθήσουμε να γεννηθεί ένας άνθρωπος είναι το καλύτερο δώρο. Και αν το προσφέρουμε αυτό δωρεάν, είναι το πρώτο και το μεγαλύτερο δώρο που μπορούμε να του προσφέρουμε. Είναι επίσης πολύ ενδιαφέρον το να εξετάσει αυτή η περίοδος της παρακολούθησης από τη ΜΕΑ, η προετοιμασία για τον τοκετό, σε ποιο βαθμό μειώνει το ποσοστό ή τον αριθμό, αν θέλετε, τοκετού σε ανωνυμία. Στατιστικά θα ήταν ενδιαφέρον να γνωρίζουμε τα στοιχεία αυτά. Στη Γερμανία υπάρχει επίσης άλλο ε, παράδειγμα παρακολούθησης της γυναίκας και της οικογένειας που περιμένει ένα παιδί ή που έχει παιδί μικρή ηλικία και που αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες. Την παρακολουθεί λοιπόν την ε, γυναίκα μία μέα και πριν από τον ε, το κετό και μετά και μάλιστα είναι ένα ζήτημα το οποίο παρακολουθούν, μελετούν πανεπιστήμια, μεταξύ των οποίων και το Πανεπιστήμιο τη Χαϊδελβέργης. Και το παράδειγμα αυτό των Γερμανίδων ΜΕΟΝ, μάλιστα πρόκειται για ένα σχέδιο του Υπουργείου, του κρατηδίου, και θα παρουσιάσουμε τις προτάσεις αυτές για την προστασία της μητέρας και του παιδιού στις 25 Μαρτίου στο Στρασβούργο. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με τον τοκετό σε συνθήκες ανωνυμίας. Πρόκειται όμως για περίθαλψη, για παρακολούθηση των δύσκολων καταστάσεων που μπορεί να αντιμετωπίσει μια μητέρα από μια μέα. Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ και σε ένα άλλο ζήτημα για το αν μπορεί να επιβληθεί ευρωπαϊκή νομοθεσία στο θέμα αυτό. Ας μην αυταπατώμεθα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν μπορούμε να νομοθετήσουμε. Νομοθετική βάση, νομική βάση δεν υπάρχει. Αυτό που θα μπορούσαμε να πράξουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι θέματα της δημόσιας υγείας να τα ρυθμίσουμε και εγώ πιστεύω ότι το να μειωθεί το κόστος ενός τοκετού σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι ένα ζήτημα με το οποίο μπορούμε να ασχοληθούμε. αλλά το να νομοθετήσουμε για την εισαγωγή του τοκετού σε συνθήκες ανωνυμίας είναι νομίζω αυταπάτητο να το επιδιώκουμε. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Παραγωτοπούλου, κυρία Κελέχ. Θα ήθελα να απαντήσω στην ερώτηση αυτή και να πω ότι στη Γαλλία δεν αναλαμβάνει την παρακολούθηση ή την διεξαγωγή του τοκετού ημέα αποκλειστικά. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα σύστημα κοινωνικής πρόνοιας για το παιδί και με ένα συμβούλιο, Εθνικό Συμβούλιο Πρόσβασης στα στοιχεία της οικογένειας. Τώρα το να βοηθήσουμε μια γυναίκα στο τοκετό μπορεί να εμφανιστεί με διαφορετικέ μορφέ. Μπορεί να έχουμε μια γυναίκα η οποία θα έρθει έγκυο ακόμη, οπότε μπορούμε ακόμη να ε, τη βοηθήσουμε, να την παρακολουθήσουμε, να τη προσφέρουμε ολόκληρο το πλέγμα ή το φάσμα βοήθεια που θα μπορούσαμε να έχουμε στη θέση μα για να τη βοηθήσουμε και να κρατήσει το παιδί, ή αν δεν αρκεί αυτό, μπορούμε να τη προτείνουμε τη δυνατότητα για το και τόσε συνθήκε ανωνυμία. Επίση, έχουμε την περίπτωση τη γυναίκα η οποία έρχεται κατευθείαν ετοιμόγενη γεννά το παιδί της και αποχωρεί αμέσως. Γιατί οι συνθήκες τις οποίες αντιμετωπίζει είναι τόσο ιδιαίτερες. Ένα παράδειγμα. Πριν από μερικά χρόνια μας τηλεφώνησε μια γυναίκα και λέει μπορεί κανείς να κάνει το κετό όταν έχει ήδη υποστεί κεσαρική τομή. Η απάντηση από τη ΜΕΑ ήταν όχι είναι επικίνδυνο κάτι τέτοιο, μια κεσαρική ακολουθεί μια άλλη κεσαρική. Δεν μπορεί να γίνει το κετός μετά από κεσαρική. Το απόγευμα λοιπόν το ίδιο εμφανίστηκε μια γυναίκα στο κέντρο μας ε, η οποία μας λέει έχω κάνει δύο ε, κεσαρικές ήδη, έχω δύο παιδιά, ο άντρας μου με έχει κακοποιήσει, επανήλθε στο σπίτι, με βίασε, δεν είχα καταλάβει καν ότι είμαι έγκυος, μόλις πρόσφατα κατάλαβα ότι κυοφορώ και μάλλον είμαι και ετοιμόγενε». Την είδαμε λοιπόν αμέσως, την εξετάσαμε αμέσως, την αναλάβαμε. Έγινε η κεσαρική, ε, με όλες βέβαια τις ιατρικές εξετάσεις, υπέρηχους κτλ. Έγινε η κεσαρική μια Παρασκευή βράδυ. Εγκατέλειψε το παιδί της. Κυριακή απόγευμα πήρε το αυτοκίνητο και γύρισε στην περιοχή στην οποία μένει, γιατί δεν ήταν κοντά σε μας. Δεν ήταν στο νοσοκομείο μου, δηλαδή το, κοντά το σπίτι της. Ε, βλέπετε λοιπόν ποιε είναι οι συνθήκε που μπορούν να οδηγήσουν μια γυναίκα. Μάλλον τελευταία στιγμή σκέφτηκε ότι αν γεννήσει μόνη τη και ενδεχομένω σκοτώσει και το παιδί, κινδυνεύει να πεθάνει, επειδή έχει ήδη περάσει δύο κεσαρικέ. Και βέβαια, ίσω να σκέφτηκε και ποιο θα φροντίσει τα δύο τη άλλα παιδιά. Όλα αυτά λοιπόν είναι συνθήκε τι οποίε πρέπει κανεί να λάβει υπόψη. Τα πάντα συμβαίνουν σε αυτόν τον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ. Θα θέλατε και εσείς να κάνετε δύο σχόλια. Πολύ σύντομα. για το θέμα του πώς μπορεί να στιγματιστεί μια γυναίκα εάν έχει υποστεί άμβλωση. Και αυτό συμβαίνει βέβαια, αλλά περισσότερο όταν έχει γεννήσει παιδί, γιατί είναι διαφορετικό το να έχει κανείς γεννήσει ένα παιδί και να το έχει εγκαταλείψει. Είναι μια εναλλακτική <coughs> βέβαια. Είναι μια λύση απελπισίας αυτή του τοκετού σε ανωνυμία για μια γυναίκα, αλλά δεν πρέπει και να παραγνωρίσουμε τα δικαιώματα του παιδιού να μπορεί να αναζητήσει τις ρίζες του. Πρέπει να εξισορροπήσουμε, να ζυγίσουμε όλες αυτές τις συνθήκες, τα δικαιώματα, τις δυνατότητες τελικά. Όσον αφορά τα δικαιώματα του παιδιού, όντως σε αυτήν την συνθήκη αναφέρεται ρητός ότι δικαιούται την πρόσβαση στα δεδομένα που συνδέονται με την προέλευσή του, αλλά επίσης δικαιούται ε, προστασίας και έχει και το δικαίωμα στην υγεία. Γι' αυτό και η γαλλική λύση στο πρόβλημα ήταν το να εξασφαλίσει την προστασία της μητέρας και του ανηλίκου και επίσης να φροντίσει τον ανήλικο διότι ε, κάποια γυναίκα τόσο νέα ε, το να γεννάει υπό μυστικότητα ε, αυτό οδηγεί σε πάρα πολύ ψηλά ποσοστά παιδικής νησιμότητας και άρα είναι πάρα πολύ σημαντική υπόθεση προστασία της μητέρας. Σας ευχαριστώ λοιπόν Ακριβώς την ίδια το ίδιο πνεύμα έχει και η δική μας νομοθεσία. Δεν βλέπω να θέλει άλλος τον ε, λόγο. Δεν υπάρχει άλλη ερώτηση. Οπότε και με τη σειρά μου θα πρέπει να ευχαριστήσω τις προσκεκλημένες μας κύριε Μαράτου και την κυρία Κέλλερ οι οποίες μας εξέθεσαν τις, παρουσίες, τις απόψεις τους μας ε, πρόσφεραν την εμπειρία τους γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική υπόθεση να υπάρχει εμπειρία σχετικά με αυτό το οποίο συζητούμε. Μιλούμε τώρα για την τύχη ενός παιδιού, την τύχη μιας γυναίκας και κάθε περίπτωση είναι μοναδική, επομένως θα πρέπει να πειστε με σοβαρότητα και με σωστή προσέγγιση ή δυνατόν. Ούτως ώστε να μπορέσουμε να ανασχέσουμε κάθε απειλή είτε για τη ζωή είτε κάποιο άλλη βλάβη της οικίας και θα πρέπει επομένω να πιέσουμε τον νομοθέτη στις χώρες μας να ε, θεσπίσουν κάποια μέτρα ούτω ώστε να πλαισιωθεί και αυτή η περίπτωση άρα θα πρέπει να έρθουμε σε με τα εθνικά κοινοβούλια και να μπορέσουμε να πετύχουμε τη θέσπιση τέτοια νομοθεσία. Κύριε Μπράγερ, σα ευχαριστούμε για την ιδέα σα για αυτήν την συζήτηση στην Επιτροπή μας. Νομίζω ότι εδώ πέρα έχουμε ένα ολόκληρο μοσαϊκό και είναι μόνο μια ψηφίδα το ζήτημα αυτών των γεννήσεων. Όλους σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας και εδώ κλείνει η συνεδρίασή μας για το πρωί θα αρχίσουμε ξανά στις 3 η ώρα και θα αρχίσουμε με ψηφοφορίες παρακαλώ φέρτε τις ηλεκτρονικές κάρτες ψηφοφορίας μην ξεχάσετε να τις πάρετε παρακαλώ και όσοι συνεργάτες βουλευτών βρίσκονται εδώ, χωρί βουλευτές, να τους το επενθυμίσουν να φέρουν το απόγευμα τις κάρτες ψηφοφορίας. Καλή όρεξη.